Καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε λίγα λεπτά για να προλάβουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να έρθουν, αλλά πήγε 9 και 10 να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης αυτής. Έχουμε επιφέρει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μας θα ξεκινήσουμε με τη συζήτηση κάποιων αναφορών, παρουσία των αναφερόντων, με την παρουσία της, συγκεκριμένα των την αναφορών 4, 5 και 6. Έπειτα έχουμε τις εκθέσεις Βάλιαν και Γκέριγκερ, η πρώτη για το πρόγραμμα δικαιωμάτων των πολιτών και η δεύτερη για την ετήσια έκθεση ελέγχου του κοινοτικού δικαίου. θα κλείσουμε την πρωινή συνεδρίαση με τη συζήτηση για την διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο και στη Ρουμανία. Μετά θα έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών και έτσι θα κλείσει το πρωινό. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε παρουσία του Επιτρόπου Σεφκοβίτς και εκεί θα γίνει μια αναδιάρθρωση του προγράμματος της ψηφοφορίας οι οποίε θα γίνουν αμέσω μετά τη συζήτηση της αναφοράς 15. Αναφορά του κυρίου Σαλτίνη σχετικά με τα απόβλητα στο Κορκόλε. Οι υπόλοιπε αναφορές θα συζητηθούν στις 19 Ιουνίου. Ιδίως ε, για τη συμφωνία άκτα επειδή ακριβώς οι αναφέροντες δεν μπορούν να παρευρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση. Η συζήτηση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Μεταξύ άλλων, για την αναφορά υπαριθμών 17 θα παρευρεθούν και τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας της Βουλγαρίας. Σε ό,τι αφορά τα παρατήματα, στο Β έχουμε αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής απάντησης της Επιτροπής Οπότε θα διτηρήσουμε αυτή την πρόταση απαράλλακτη, όπως έχει μοιραστεί στους συναδέλφους, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Να επισημάνω στους συναδέλφους ότι η κυρία Ντεμπρούν παρατήθηκε από τη θέση της στο Ευρωκοινοβούλιο για λόγους υγείας. Ήταν ε, μέλος της Επιτροπής μας και συντονίστρια εδώ η κυρία Ντεμπρούν, αλλά εγκατέλειψε το αξιωμά και της αποστέλω ευχές, νομίζω ευχές από όλους μας, που θα φροντίσω να τις διαβιβαστούν τις ερχόμενες ημέρες για την υγεία της. Σας ζητώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι είναι εγκεκριμένη. Ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο σημείο, δηλαδή την πρώτη αναφορά υπαριθμών 4 στην Εμερήσια διάταξη, αναφορά του κυρίου Κριστόμπαλα Γκουαντολάθα, ισπανική Ιθαγένεια, εξ ονόματο του Γεωργικού Συνεταιρισμού Ασάγια. Να του δώσω ευθύ αμέσω το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ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 Εκτός από τον περιορισμό των σημείων εισόδου, θα προτείναμε επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ε, γραφείου που θα είχε ε, αυτές τις αρμοδιότητες. Και όσον αφορά στην αμοιβαιότητα, όσον αφορά δηλαδή ε, την διατήρηση των, της ανοχής ε, κατά την εισαγωγή. Είναι αλήθεια ότι στις τρίτες χώρες υπάρχει μια απαγόρευση στις εισαγωγές ε, για προϊόντα που, ε, στα οποία έχουν εφαρμοστεί κάποιες ουσίες που είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αντίφαση γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διεθνή συμφωνία αναφορικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε να γίνει μια ξεκάθαρη συμφωνία με το αντίστοιχο διεθνές ε, ε, ε, σώμα, τον, FAO, τον, τον ΠΟΗ, τον FAO. Έτσι λοιπόν, όταν μία συγκεκριμένη χώρα καταθέτει αίτηση για μία ανοχή, να απαιτείται ακριβώς να απαιτούνται ακριβώ τα ίδια έγγραφα που υπάρχουν, που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν θα πρέπει να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι ε, καταναλωτές να μπορούν να εμπιστεύονται τα προϊόντα διότι αυτά θα σέβονται κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που είναι πολύ ε, αυστηροί. Εφόσον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους πιο περιοριστικούς κανόνες για τη φυτοπροστασία στον πλανήτη, οι Ευρωπαίοι αγρότες είναι ε, υπόκεινται σε αθέμητο ανταγωνισμό. Όλα αυτά για να εγγυηθούν την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών και οποιασδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ε. Σας ευχαριστώ. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. κύριος Ντράκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο πρώτο τμήμα της αναφοράς είχαμε δώσει μια γραπτή απάντηση για το πρώτο τμήμα της αναφοράς αλλά αντί να σας τη διαβάσω, θα ήθελα να τη σχολιάσω. Να σχολιάσω μάλλον αυτά που μόλις είπε ο αναφέρον. Ότι δεν έχει η Κομισιόν ε, αρκετά μέτρα για ένα πακέτο ζυζανιοκτώνων τα οποία θα είναι επαρκή να, ώστε να εμποδίζεται η ανθεκτικότητα, η δημιουργία ανθεκτικότητας των φυτών. Έχουμε κάποιους κανόνες για την εισαγωγή νέων ζυζανιοκτώνων και κάθε χρόνο φαίνεται ότι υπάρχουν νέα ζυζανιοκτώνα τα οποία ε, κατατίθεται ε, για αξιολόγηση. Αυτή είναι δηλαδή μια συνεχής διαδικασία. οι κατασκευαστές ε, των φυτοφαρμάκων που πρέπει να καταθέσουν ένα ντοσιέ είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι η Κομισιόν ε, που τα παράγει. Έχει μόνο το καθήκον της αξιολόγησης. Η ΕΦΣΑ κάνει την ε, εκτίμηση κινδύνων, όπως αναφέρατε, για το περιβάλλον συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα για την υγεία των καταναλωτών ε, και ε, οι αξιολογήσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η Κομισιόν είναι τέτοια ώστε ε, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται να είναι ασφαλή. Δηλαδή αυτά που δεν έχουν αρκετά στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλή είτε για τους καταναλωτές είτε για το περιβάλλον ε, δεν ε, συνεχίζουν να απολούνται. Αυτό χωρίς ε, να θίγονται τα συμφέροντα ή ουδήποτε εκ των ενδιαφερομένων, είτε δηλαδή αυτού που πουλάει είτε του καταναλωτή. Δεν είναι ότι απαγορεύουμε δηλαδή τελείως τη χρήση των φυτοφαρμάκων, αλλά τα χρησιμοποιούμε υπό αυστηρούς κανόνες. Έτσι λοιπόν αυτοί που ενδιαφέρονται ε, να περάσουν ε, ε, μια έγκριση για ένα φυτοφάρμακο θα πρέπει να καταθέσουν αρκετά στοιχεία έτσι ώστε να, να επιτραπεί στους χρήστες να καταχωρήσουν αυτά τα φυτοφάρμακα για τους σκοπούς που μόλις ανέφερε ο αναφέρον. Άρα δεν απαγορεύει η Κομισιόν, αλλά ε, στην ουσία επιτρέπει τη χρήση. Επίσης, μας ανησυχεί το γεγονός της δημιουργίας ανθεκτικότητας σε, συγκεκριμένα ζυζάνια. Σε, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε κάποιες είναι πιο ανησυχητική περίπτωση, υπάρχει ένα πακέτο ε, ουσιών για, την ίδια, για τον ίδιο συνδυασμό ε, ζυζανίων. Παρασύντων. Υπάρχει λοιπόν ένα επαρκές ε, πακέτο για τον έλεγχο των ε, παρασύτων με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα. Τώρα για την ανοχή κατά την εισαγωγή. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι ως προς αυτό το θέμα της ανοχής κατά την εισαγωγή στην Κομπισιόν, γιατί ε, η, η ανησυχία του, λοιπόν, του αναφέροντος είναι και δική μας ανησυχία. Δεν επιτρέπουμε Τέλος πάντων, οι κανόνες είναι τέτοιοι ώστε οι χρήστες ή οι ετούντες για υπολείμματα, ε, δηλαδή μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, NL, ε, ε, να ε, πληρούν τους κανόνες μας. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξουμε ε, τα ζυζανιοκτώνα χρειαζόμαστε αυτές τις, αυτούς τους κανόνες ανοχής κατά την εισαγωγή. Για τη διόρθωσή τους οι κανόνες είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται για χρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτά τα όρια. Ε, έτσι λοιπόν θέλουμε κατά την αξιολόγηση να γίνονται σεβαστοί αυτοί οι κανόνες. Από την άλλη, μπορεί να φαίνεται και ίσως να είναι και η άποψη από, η οποία ανέπνευσε τον αναφέροντα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά τέτοια ε, όρια για ουσίες οι οποίες έχουν αποσυρθεί από την αγορά, δεν έχουν ε, καταργηθεί. Ε, έχουν αποσυρθεί γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των ε, κατασκευαστών, των καλλιεργητών κτλ. Δεν έγινε κάποια κατάθεση λοιπόν στην Κομισιόν. Έτσι λοιπόν πολλές ουσίες έχουν αποσυρθεί από την αγορά και υπάρχουν MRLs για πολλά ΑΟΚ δηλαδή, για πολλά ε, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για άλλα ε, τα οποία ε, έχουν σταματήσει να έχουν άδεια. Ε, βλέπουμε τελικά ότι ακόμα και τρία χρόνια μετά την αναστολή της χρήσης τους ε, παραμένουν υπολείμματα αυτών των ουσιών ε, σε πολλά τρόφιμα. Δηλαδή για πάνω από 18 μήνες ε, συνεχίζει η χρήση τους και μετά χρειάζεται άλλους 18 μήνες έτσι ώστε να ελεγχθούν τα όρια. Από την άλλη, χρειάζονται γύρω στα 10 χρόνια για να φύγουν τελείω από την διατροφική αλυσίδα. Υπάρχει λοιπόν κάποιος λόγος που διατηρούμε αυτά τα ανώτατα όρια καταλήπων. Είναι αλήθεια επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις που επιτρέπουμε αυτά τα τα όρια καταλήπων, τα MRL, ε, για ουσίες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όμως είναι πάρα πολύ ε, σπάνιες και βασίζονται στον κόντεξ αλιμεντάριους, διεθνεί κανόνες ή από άλλους κανόνες ε, του ΠΟΕ, το, από το SPS. Και είμαστε επιφυλακτικοί ε, ως προς την προς το να επιτρέψουμε τέτοιες ε, ε, ουσίες για τρίτες χώρες. Και οι εξαιρέσει ε, ουσιαστικά δόθηκαν σε χώρες όπως η Νότιο Αφρική, αλλά διασφαλίζουμε πάντοτε ότι αυτές οι εξαιρέσεις που μας επιβάλλει ο και ο Κόντεξ διασφαλίζουμε ότι οι αρχές στη Νότιο Αφρική γνωρίζουν ότι είναι όλο αυτό προσωρινό και θα βγάλουν αυτές τις ουσίες από την αγορά. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρατε περιβαλλοντικούς ε, λόγους ε, για την απόσυρση μιας ουσίας από την αγορά. Οι κανόνες για το περιβάλλον ε, είναι κανόνες που έχουμε εμείς και δεν μπορούμε να τι επιβάλλουμε στις τρίτε χώρες και δεν είναι αναγνωρίσιμοι και από τον ΠΟΕ. Οι κανόνες ε, για τους ετούντες ε, φυτοφαρμάκων, α πούμε, ε, είναι ε, κανόνες ε, που αφορούν και τους καταναλωτές στην Αφρική, στην Κίνα και έτσι μέσα από τις συνθήκες μας και τις επαφές μας προειδοποιούμε γι' αυτό. Στη, Σαγκάνη, στη Σαγκάη πριν από λίγες ημέρες είχαμε την Επιτροπή του Κόντεξ Ελμετάριους για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και προειδοποιήσαμε τις αντιπροσωπείες σχετικά με το αν υπάρχουν ανησυχίες για κάποιες ε, ε, ουσίες και είπαμε ότι δεν θα επιτρέφουμε αυτές, αυτά τα νότατα όρια για πολύ καιρό και όταν υπάρχουν ε, νέα όρια στον κόντεξ θα είμαστε αντίθετοι και το αποτέλεσμα θα είναι να μην υιοθετηθεί γενικά αυτό το όριο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμμετάσχει και ο εκπρόσωπο ε, τη Γενική Διεθνή Άγκρη, ο κ. Δεμπέκερ. Είναι στην αίθουσα. Μάλιστα. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Είμαστε βέβαια σε στενή επαφή με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Καταναλωτών. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της αναφοράς είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαραίτητα προϊόντα για να προστατεύουν τις σοδιές αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μην παραβλέπεται η ανάγκη εξασφάλισης βιωσιμότητα στη γεωργία. Και υπάρχουν και διεθνείς υποχρώσεις, που, από τις οποίες δεν μπορούμε να αποφύγουμε Έχει σημασία λοιπόν, έχουν σημασία και οι σχέσεις μας με τους εταίρους μας σε τρίτες χώρες και βέβαια και να υποφεληθεί και από αυτές αλλά και από την Ευρωπαϊκή Γεωργία και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Ευχαριστούμε. Το ρόλο έχει γυρίζει η κυρία Χέρνης Καρσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απήντησε στους αναφέροντες γραπτός στο έγγραφο αυτό η απάντηση χωρίζεται σε τρία μέρη. Πρώτα απ' όλα η συντόμευση της ε, ταχείας διαδικασίας για την έγκριση δραστικών ουσιών. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι προκειμένου να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της γεωργίας και την προστασία των καλλιεργειών ορίζονται ελάχιστα όρια για δραστικές ουσίες. Αυτό όμω θα το περιμέναμε από την Επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβριο, πριν από ένα εξάμεινο. Επί ένα εξάμεινο τουλάχιστον, ο αναφέρον ακριβώς ε, καταγγέλει την απουσία τέτοιας ρύθμισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπέβαλε έγγραφο που να αναφέρουν αυτές τις προδιαγραφές, τις, έκτακτες, τις με φυτογειονομικά μέτρα. Θα έπρεπε λοιπόν ένα φορά να γίνει δεκτή και να βρεθεί κάποια λύση. Παράταση δηλαδή της χρήσης των δραστικών ουσιών. Επαναλαμβάνω λοιπόν, από τις 14 Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε ήδη να μας έχει υποβάλει αυτό το έγγραφο, πράγμα που δεν έγινε. Το έγγραφο δεν υπευλήθη και θα έπρεπε να έχει συζητηθεί ώστε το νομοθετικό μας έργο να έχει επιτελεστεί εγκαίρως. Όχι όταν ε, αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει χρόνο να μας το στείλει. Έπειτα, για τις ασθένειες, τις νόσους και τους πολεμικούς οργανισμούς που προέρχονται από τρίτες ε, χώρε. Μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εδώ υπάρχει αυξητική τάση και ότι υπάρχει και σχετική διάθεση αναθεώρηση τη ε, νομοθεσία. Αυτό προβλεπόταν ήδη για την περασμένη χρονιά. Ο αναφέρον έχει συμμετάσχει στην όλη και την παρακολουθεί. Όμω δεν έχει ξεκινήσει επισήμω η όλη διαδικασία. Πώ να συμμετάσχει λοιπόν, ε, προσφέροντα τη συνεισφορά του και τι απόψει του. Εδώ λοιπόν και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθυστερήσει. Και ε, βλάπτει τα συμφέροντα του αναφέροντος. Εφόσον η νομοθετική διαδικασία λοιπόν δεν έχει ξεκινήσει, εφόσον δεν έχουν οργανωθεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λογικό είναι να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσει του αναφέροντος. Έπειτα, τρίτο στοιχείο στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας μιλάει για την ανοχή στην εισαγωγή δραστικών ουσιών που προέρχονται από τρίτες χώρες. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι κάποια φυτοπροστατευτικά μέτρα δεν γίνονται αποδεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον προέρχονται από τρίτες χώρες, ακόμη και αν σε πολλές περιπτώσεις, λέει μάλλον σε αρκετές περιπτώσεις, δεν λέει σε όλες, ακόμη και αν αυτό δεν αφορά την προστασία των καταναλωτών. Εδώ υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων επίσης. Αλλά οι συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις ε, δεν καλύπτουν ε, την περίπτωση του αναφέροντος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν επαρκεί έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τέτοια φυτοφάρμακα να μην χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Λόγω χάρη δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια συστατικά, τι ίδιε ουσίε για τα εσπεριδοειδή στη Βαλένθια τη Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Και βεβαίω οι Ευρωπαίοι καλλιεργητές θα βρεθούν να έχουν να βρίσκονται σε δυσκαιρέτερη θέση από τους Βόρειο λόγου χάρη που, δεν διαθέτουν, που διαθέτουν άλλα φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως αυτή ακριβώς η των εσπεριδοειδών. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει και το θέμα των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τρίτες χώρες ε, και πάλι για τα εσπεριδοειδή. Όταν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί θέλουν να αποστείλουν τα προϊόντα τους σε τρίτες χώρες, υπάρχουν πρωτόκολλα ιδιαίτερα αυστηρά που έχουν να κάνουν ακριβώ με την παρουσία κάποιων επιβλαβών οργανισμών ή νόσων που εμείς δεν έχουμε τρόπο να τα θεραπεύσουμε ακριβώ γιατί δεν καλύπτονται από τους καταλόγους τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει λοιπόν αμοιβαιότητα στην εισαγωγή σπυριδοειδών ε, από τρίτε χώρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μας αγγιηθεί καν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα φτάσουν ε, στην ευρωπαϊκή αγορά με τις ίδιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τα ίδια μέτρα προστασίας των καλλιεργιών. Μπορεί λοιπόν στην επικράτειά μας να βρεθούν επιβλαβείς οργανισμοί και νόσοι που δεν υπήρχαν ε, προηγουμένως ακριβώς λόγω των εισαγόμενων προϊόντων και να μην έχουμε και τα φάρμακα, τα μέτρα προστασίας ώστε να τα αντιμετωπίσουμε. Εφόσον λοιπόν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συνάδουν με τα δεδομένα που έχουμε από μελέτε, λόγω χάρη του Πανεπιστημίου Πολυμπλάν τη ε, Βαλένθια, που λέει ότι κάθε εβδομάδα έχουμε μια νέα ασθένεια που εμφανίζεται στι ε, ευρωπαϊκέ καλλιέργειε. Περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει κάπω. Αποστήλαμε επίστολη στον ε, Επίτροπο που είναι επιφορτισμένος με τα θέματα γεωργία, ακριβώ για να έχουμε μια άμεση απάντηση και περιμένουμε ακριβώ μια απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Γιατί πλήττεται το τομέα των εισπροειδευτών στην Ευρώπη. Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα. Πρόκειται πρωτίστως όχι μόνο για θέματα περιβάλλοντος αλλά και για την εξασφάλιση της προμήθειας τροφίμων και για ε, τους ανθρώπους και για τα ζώα και καθεξής. Αυτή είναι η βασική αρχή που πρέπει να διέπει όλους τους κανόνες που θα εφαρμοστούν. Δεύτερο κύριο στοιχείο είναι της εμπορίας, της διάθεσης του εμπόριου δηλαδή των προϊόντων αυτών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να παράγουν οι παραγωγή. Τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή του κόσμου. Υπάρχουν κανόνες εμπορικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από το διεθνές σύστημα και αυτοί έχουν αρνητικό, αρνητική επίπτωση. Δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται, δηλαδή με ανισότητες σε ό,τι αφορά τους ελέγχους της χρήσης των ζυζανιοκτώνων και άλλων εντομοκτώνων κλπ. στα διάφορα σημεία του πλανήτη και οι συνέπειες που, έχουν, που έχει διαθεσή του σε, όλα, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο οι Ευρωπαϊκές Αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ασκούν αυστηρούς ελέγχους και στις εισαγωγές, διότι φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Για παράδειγμα, για τα εσπεριδοειδή, όπου φαίνεται ότι η έλεγχη είναι πολύ λιγότερη αυστηρή, πολύ λιγότερο αυστηρή. Για παράδειγμα, η έλεγχη επί των εσπεριδών, επί των εσπεριδοειδών που εισάγονται από τρίτες χώρες είναι πολύ λιγότερο αυστηρή από αυτούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που προέρχονται από την Ισπανία. Εκτός τώρα από τα ζυζανιοκτώνα και τις διάφορες ενεργές ουσίες υπάρχουν και πολλές άλλες δυνατότητες για την καταπολέμηση βλαβερών εντόμων και άλλων. Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα δηλαδή προϊόντων που χρησιμοποιηθούν πολλές οικολογικές, δηλαδή βιολογικές δυνατότητες που ε, αποδίδουν. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την παραγωγή τροφίμων, αλλά αυτό εξυπηρετεί και το ίδιο το περιβάλλον. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Για όσα είπε και η συνάδελφος, πραγματικά η αναφορά αυτή πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά νομίζω πρέπει να ενημερωθεί και η Επιτροπή Γεωργία ε, του Κοινοβουλίου μα για το τι συμβαίνει, για την όλη κατάσταση που παρουσιάζει η αναφορά. Η επιστολή λοιπόν που θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποσταλεί και στον πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργία ώστε να ενημερωθούν και να μπορέσουν να ετοιμάσουν μια σχετική γνωμοδότηση, ένα σχέδιο έκθεση για το θέμα αυτό. Από ό,τι φαίνεται από τα σχόλια των συναδέλφων, τα θέματα αυτά επηρεάζουν τον τομέα στον οποίο εργάζεται ο αναφέρον και βεβαίως και άλλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη συνάδελφό μου κυρία Εράνς που παρουσίασε πλήρω το πρόβλημα, συμφωνώ και με τον μόλις προαλήσατε συνάδελφό μου, να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Νομίζω ότι και άλλες επιτροπές ενδιαφέρονται, η Νομική Επιτροπή αλλά και η Επιτροπή Εμπορίου και θα γνωμοδοτήσουν. Εδώ υπάρχει ανάγκη αναλήψεως δράσεως, διότι υπάρχουν και αντικίνητρα και στην νομοθεσία. Η Κομισιόν είπε ότι διάφορες ουσίες έχουν εξαιρεθεί. Το πρόβλημα είναι εάν ένας παραγωγός ζυζανιοκτώνων, για παράδειγμα για τα δημητριακά, και εδώ μιλούμε για εκατομμύρια εκτάρια, προχωρεί, κάνει μια διαδικασία εγκρίσεως και αυτή αποδίδει. ενώ ένας για παράδειγμα ο οποίος καλλιεργεί άνθη, λουλούδια και στη Γερμανία για παράδειγμα δεν έχουμε πολλούς τέτοιους, είναι πολύ περιορισμένη η παραγωγή. Δεν αξίζει για αυτόν να προχωρήσει σε ειδική διαδικασία, να ζητήσει δηλαδή ειδική διαδικασία εγκρίσεως παίρνει αυτό που χρησιμοποιείται για τα δημητριακά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα ειδικό προϊόν για την παραγωγή λουλουδιών. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος δηλαδή να υπάρχουν τα απαραίτητα προϊόντα και να μπορούν να εγκρίνονται με ταχύτητα και για μικρές παραγωγές. Το άλλο πρόβλημα είναι, όπως είπε σωστά η κυρία Ράνς, ότι η φύση εξελίσσεται και μας θέτει διαρκώς προ νέων προκλήσεων. Και το τρίτο πρόβλημα είναι η αλλοδαπή. Δηλαδή, η αλλοδαπή με ήττα εννοώ, όπου έχουν τελείως διαφορετικούς κανόνες, πολύ πιο χαλαρούς. Εάν, για παράδειγμα, απαγορεύεται ένα ζυζανιοκτόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντα όμως εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, κανονικά δεν θα πρέπει εδώ να υπάρχει απολύτως καμία ανοχή απέναντι σε επιβάρυνση με ζενιοκτώνα τέτοιων προϊόντων. Αυτό το χρωστάμε στους πολίτες. Δηλαδή, είτε θα πούμε ότι είναι επικίνδυνο το ζανιοκτώνο και επομένω δεν πρέπει να ανεβρίσκονται ίχνη του ή εάν επιτρέψουμε, αν επιτρέψουμε κάποιες ανοχές, τότε δεν είμαστε πλέον ειλικρινεί. Δεχόμαστε τότε ότι ε, δεν είναι και τόσο επικίνδυνο. Για μένα αυτό είναι μέγα θέμα προς συζήτηση, διότι αν επιτρέψουμε κάποιες ανοχές, το ξέρουμε άλλωστε και οι ίδιοι Κάθε χρόνο έχουμε αποκλήσεις, εξαιρέσεις για προϊόντα τρίτων χωρών. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να ελέγξει και την τελευταία ντομάτα και το τελευταίο λεμόνι. Είναι όμως πολύ σημαντικό το πρόβλημα, το οποίο έθεσαν δηλαδή οι αναφερόμενοι, γιατί πρόκειται εν τέλει για την προστασία της υγείας των ανθρώπων, αλλά και την προστασία της υγείας των φυτών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Πρόκειται όμως και για θέματα στρεβλώσεως του ανταγωνισμού. Γι' αυτό πρέπει οι αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και να κληθούν και οι άλλες συναρμόδιες επιτροπές να γνωμοδοτήσουν. Και εσείς κύριε Ράνς είστε μέλος στην Αγροτική Επιτροπή, στη Γεωργική Επιτροπή και εγώ να ζητήσουμε λοιπόν η Επιτροπή Γεωργίας να εγκύψει εντατικά στο πρόβλημα. Δεν ζητούν άλλοι συνάδελφοι το λόγο, οπότε να δώσω το λόγο πάλι στον αναφέροντα για να απαντήσει. <clears throat> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ρύζι είναι ένα φυτό το οποίο χρειάζεται τέσσερις μήνες ε, για την παραγωγή του. Είπαμε πριν από λίγο ότι έχουμε μια θεραπεία για μια συγκεκριμένη ε, ασθένεια, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, τέσσερις διαφορετικές θεραπείες γιατί υπάρχει η ανθεκτικότητα σε κάποια προϊόντα. Δεύτερον, Υπάρχει και η έγκριση για τις ε, ε, ελάσσον ίσονος χρήσης προϊόντα. Στην Ισπανία κάθε χρόνο έχουμε εκατοντάδες προϊόντα για τα οποία ε, ζητούμε να υπάρξει μια εξαιρετική άδεια, καταξαίρεση δηλαδή. Το καταλαβαίνω αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο κόντεξ ε, όμως ε, το να ε, εξάγουμε μανταρίνια στι ε, στις ΗΠΑ μπορεί να, έχει ένα, να υπόκειται σε ένα πρωτόκολλο, αλλά όταν έρχονται οι δικοί μας, οι Αμερικανοί, έρχονται στα δικά μας εργοστάσια και βλέπουν ακριβώς τι συμβαίνει μέχρι να φτάσει να διαμετακομιστεί ένα προϊόν στο αμερικανικό ε, λιμάνι ε, και να εγκρίνουν ε, μόνο συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία έχουν άδειε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Έχουμε εξαιρετικό κόστος για κάθε εξαγωγή μας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έτσι λοιπόν όταν εισάγουμε σε επίπεδο ΑΟΚ, εάν ένα προϊόν δεν έχει έγκριση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο ανώτατο όριο ε, για τις εισαγωγές, ε, το οποίο ε, θα αφορά και όσα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό. Για να φτάσουμε στο συμπέρασμα, θεωρώ ότι ε, τους τελευταίους μήνες οι γεωργοί έχουν ε, πρόβλημα με νέα παράσιτα. Έχουμε όλο και λιγότερα προϊόντα που αντιμετωπίζουν αυτά τα παράσια, παράσιτα, ειδικότερα ε, στην Μεσόγειο, όπου υπάρχει παγκοσμιοποίηση και των παρασίτων. Ζητώ λοιπόν από την ε, Πρόεδρο να κάνει ό,τι γίνεται με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Ε, χρειαζόμαστε ασφάλεια. Είμαστε εμείς οι γεωργοί αυτοί που χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα και τέλος πάντων πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστική τιμή ε, και αν πρέπει να επαναλαμβάνουμε την θεραπεία λόγω έλλειψης προϊόντων είναι μεγάλο το κόστος. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι και ιδιαίτερα επίκαιρο και ευαίσθητο. Και βλέπω και πώ απασχολεί τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ομόφωνη η απέτηση των συναδέλφων να γύρουμε το θέμα αυτό και στι υπόλοιπε αρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Και πολύ σωστά μα είπε και ο Εμμανό συνάδελφο ότι όχι απλώς θα πρέπει να ζητήσουμε γνωμοδότηση από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές, αλλά και να ενεργοποιηθούν διότι το θέμα που μας απασχολεί θα πρέπει να επιληθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα κιόλας. Ε, νομίζω δεν υπήρξαν αντορίσεις ως προς αυτό. Συμμερίζομαι και την απέτηση της συναντέλφου Γκαρσία να απευθυνθούμε και στον αρμόδιο επίτροπο και να ζητήσουμε από τους εκπροσώπους της Επιτροπής κάτι παραπάνω από αυτά που μας απέστειλαν γραπτός. και από όσα μας είπαν σήμερα οι εκπρόσωποι των δύο γενικών διευθύνσεων. Νομίζω λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να παραμένει ανοιχτή η δικασία της αναφοράς αυτής, όπως ζήτησαν όλοι οι παρεμβαίνοντες. Σας ευχαριστώ και πάλι και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Η αναφορά υπαριθμών 5, η οποία έχει υποβληθεί από ομάδα Ισπανών πολιτών με όνομα Πλαταφόρμα από la Defensa de los Valles Verdes, για την προστασία, πλατφόρμα δηλαδή για την προστασία των ε, πράσινων παιδιάδων. Εξ ονόματος του κυρίου Γαρβεσφία, λοιπόν, θα του δώσω το λόγο για πέντε λεπτών. και πέντε λεπτά. Είναι εδώ, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς και την Επιτροπή που μας δίδεται άλλη μια ευκαιρία να μιλήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντως, στις 28 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Αναφορών μπορέσαμε να σας ε, παραθέσουμε την κατάσταση σε ένα ε, θέμα μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας για την Ισπανία. Ζητήσαμε να ληφθούν μέτρα επιγόντως και θέλαμε οι ευρωπαϊκές και οι ισπανικές ε, αρχές ε, να ολοκληρώσουν και να σταματήσουν αυτό που εμείς θεωρούσαμε μια επίθεση σε μια ιδιαίτερου κάλουσα περιοχή. Μετά από τέσσερις μήνες δυστυχώς συνεχίζουμε με τα ίδια επιχειρήματα να ε, πείσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές ε, να επομιστούν το βάρος ε, των ευθυνών τους, γιατί είναι οι θεματοφύλακες του ευρωπαϊκού νόμου και πρέπει να πείθουν τον κόσμο να σέβεται την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχω τρία σημεία που θέλουν να φτιάξουν μια γενική εικόνα για την αναφορά μας. Καταρχάς, αυτό που είναι κατάφορη περιβαλλοντική ζημιά σε μία ε, ζώνη ειδική προστασίας που προστατεύεται από την Επιτροπή, ε, σύμφωνα με την έκθεση της ε, Κομισιόν της 27ης Ιανουαρίου, που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες από τις Ισπανικές Αρχές, σύμφωνα με τις οποίες ε, δεν υπάρχουν ε, ε, ζημιά, δεν υπάρχει ζημιά στον υδροφόνορο ορίζοντα, ότι το ποσό της γεώτρησης, η ποσότητα της γεώτρησης είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη διαθέσιμη ποσότητα. Η έκθεση των Ισπανών βασίζεται σε μια έκθεση του Γεωλογικού και Ινστιτούτου και Ινστιτούτου Εξορίξεων στην Ισπανία. δεν, δεν αμφισβητούμε εμείς την εγκυρότητα αυτού του Ινστιτούτου. Όμως η σημασία και η ποιότητα ε, της έκθεσης ε, του Διευθυντή του Εθνικού Πάρκου, που είναι δηλαδή το ύψιστο δυνατό επίπεδο ε, και την οποία καταθέσαμε ως επιπλέον τεκμήρια για να υποστηρίξουμε την αναφορά μας τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο, ε, ένα Εγγραφά 11 σελίδων που δείχνει ότι υπάρχει πολύ σημαντική περιβαλλοντική ζημιά, ξύρανση των πηγών και ε, όλο αυτό έχει να κάνει με όλα αυτά τα μέσα συλλογής υδάτων που μαζικά ε, κάνουν γεωτρήσεις ε, σε ένα δίκτυο της Natura 2000. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτά τα στοιχεία λοιπόν που μας έχει δώσει η ύψιστη αρχή του φυσικού πάρκου αυτού. Επίσης, ε, μας ζητήθηκε να ε, δούμε το άρθρο 12 της ε, οδηγίας που λέει ότι ε, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στις αρχές και να ζητήσει να αναλυφθεί δράση. Εμείς το κάναμε αυτό κυρία Πρόεδρε, ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές στην Ισπανία και από τότε ήρθαμε και σε επαφή με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταθέσαμε τεκμήρια και δεδομένα και ο διευθυντής του Φυσικού Πάρκου πήγε και αυτό στις ε, ε, εθνικές αρχές μας ε, με βάση το ίδιο άρθρο για να ζητήσει από αυτές να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και να συμμορφωθούν με την οδηγία για το περιβάλλον. Το τρίτο σημείο είναι το πιο δύσκολο. Παρά τα όσα εξήγησα, συνεχίζει αυτή η μαζική συλλογή υδάτων ε, σε αυτή την ε, ε, περιοχή ειδική φυσικής ομορφιάς, φυσικού κάλους. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί, αυτές οι εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν να βλάπτουν το περιβάλλον ανεπανόρθωτα και οι εθνικές αρχές ακόμη δεν έχουν λάβει μέτρα όχι μόνο επίγοντα μέτρα, αλλά άμεσα μέτρα. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Ε, γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας, για να σας θυμίσω τα διάφορα στοιχεία να σας ε, επαναλάβω τα επιχειρήματα του Διευθυντή του Φυσικού Πάρκου ε, που λένε ότι πρόκειται για μία κατάφορη μη συμμόρφωση με την ε, οδηγία για το απτινά και για, την, και για το περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι ως θεματοφύλακες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να κάνουν κάτι, πρέπει να αναλάβουν δράση για να αποφύγουν ε, αυτό που ε, δημιουργεί ένα επανόρθωτη ζημιά. Οι ευρωπαίοι πολίτες ε, έχουν συμφέρον. Πρέπει να εργαζόμαστε με βάση την αρχή της, πρόληψης που είναι ο βασικός πυλώνας της περιβαλλοντικής πολιτικής μας. Υπάρχουν άνθρωποι στα ευρωπαϊκά όργανα ε, που ε, αποποιούνται των ευθυνών τους. Και το ίδιο γίνεται και με τις ισπανικές αρχές, ε, οι οποίες επιτρέπουν την βλάβη στο περιβάλλον σε μια ιδιαίτερο κάλους περιοχή. Αυτή λοιπόν η παραβίαση, η μη συμμόρφωση είναι κάτι συστηματικό Παρόμοια, περιπτώση, παρόμοια περίπτωση είχαμε στο παρελθόν. Ε, αν είχε γίνει ε, κάτι ε, στην, στις περιπτώσεις Ντονάνια και Μέλ, για παράδειγμα, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Μαρτίν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, είπε ο Επίτροπος σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή αυτή... εξετάζει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το σύστημα αυτό αρδεύσεως με νερό που θα αντλείται από το Εθνικό Πάρκο Καθόρονα και που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ειδικής προστασίας για την προστασία των πτηνών και είναι και τμήμα ε, ευρύτερου χώρου προστασίας Natura 2000. Ο αναφερόμενος πρόσθεσε διάφορα στοιχεία. Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την ικανότητά μας αναλύσεως όλων των ε, δεδομένων. η αναφορά ισχυρίζεται ότι δεν συμμορφούνται το έργο με τις οικίες οδηγίες, οδηγία πλαίσιο για τα νερά και άλλες. Τρεις φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε στις Ισπανικές Αρχές σε μια προσπάθεια να διευκρινίσει την μελέτη επιπτώσεων του έργου την ζημιά που ενδέχεται να επιφέρει δηλαδή στη, στους ειδικά προστατευόμενους αυτούς βιοτόπους. Καθώς επίσης και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα αυτή αυτή ύδατος που θα κατασκευαστούν. Η Κομισιόν σήμερα δεν είναι σε θέση να είναι βεβαία για το εάν όντως παραβιάζονται οι σχετικές οδηγίες. Λόγω της απουσίας των ε, πληροφοριακών στοιχείων που ανέφερα προηγουμένως, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την ανάλυση των δεχομένων αρνητικών επιπτώσεων. Στη βάση των πληροφοριών που διαθέτουμε φαίνεται ότι οι Ισπανικές αρχές που είναι αρμόδιες για την διαχείριση του τόπου αυτού αναγνωρίζουν ότι ίσως υπάρξουν αρνητικέ επιπτώσεις από την κατασκευή των ταμιευτήρων. Θα αρχίσω λοιπόν με την τελευταία οδηγία που αναφέρει ο αναφερόμενος στην αναφορά του. Το άρθρο 12 της οδηγίας καταστρώνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θεμελιώνει εύλογα δικαίωμα να του επιτρέπει να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές λόγω του, της επαπειλούμενης, των επαπειλουμένων μάλλον κινδύνων να αναστείλουν τα μέτρα. Στην οδηγία προβλέπεται μηχανισμός που εξηγεί πώς υποβάλλονται οι σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές. Και επιτρέπει επίσης στα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν ισχυρισμούς. Η αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους σχετικά με την απόφασή της και αιτιολογημένα δηλαδή, εάν θα δεχθεί ή όχι τις ενστάσεις αυτές. Το άρθρο 13 λέει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από ανεξάρτητο όργανο ή από δικαστήριο να εξετάσουν την νομιμότητα των αποφάσεων της διοικήσεως. Δεδομένων και των διατάξεων του Εθνικού Νόμου υπάρχει και η δυνατότητα επιδίκασης αποζημίωσης. Βέβαια, είναι απαραίτητο πρώτα να εξαντληθούν οι διοικητικές διαδικασίες πριν να καταλήξει η υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου. Στη βάση των πληροφοριών που διαθέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση να πούμε με σιγουριά ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των αναφερομένων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει και να διερευνήσει τους ισχυρισμούς περί αρνητικών επιπτώσεων. Για τις άλλες οδηγίες τώρα που αναφέρονται στην αναφορά, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, η οδηγία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Φαίνεται πως το έργο, του έργου μάλλον έχει προηγηθεί η μελέτη επιπτώσεων. Είναι σημαντικές διατάξεις αυτές βέβαια στην οδηγία. Όπως ορισμένες διατάξεις, όπως η καθυστέρηση δημοσιεύσεως από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές της Ανδολουσίας, αυτό όμως είναι ενδεχόμενο θέμα παραβιάσεως του εθνικού δικαίου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν εύλογε αμφιβολίες σχετικά με την πλήρη τήρηση των διατάξεων τη οδηγία, διότι στην βάση των πληροφοριών που διαθέτουμε είναι αδύνατο να μην λάβουμε υπόψη το ενδεχόμενο να μην έχουν γίνει σωστά οι μελέτε των επιπτώσεων και ιδίως της απειλή κατά φυτών και έμβιων όντων. Επίσης δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις. Τώρα για την οδηγία περί βιοτόπων. Οι ισπανικές αρχές, όπως είπα πριν, δεν έχουν ακόμη μπορέσει να διαπιστώσουν ότι έγινε επαρκής μελέτη επιπτώσεων για τα ενδεχόμενα, τις ενδεχόμενων μάλλον επιπτώσεων της κατασκευής των ταμιευτήρων αυτών υδάτος στο περιβάλλον της περιοχής. Εκτός από αυτό, φαίνεται πως λόγω της αρδεύσεως από τον υδροφόρο ορίζοντα, λόγω τη αντλήσεω μάλλον υδάτων, ενδέχεται να υπάρχει και εκεί αρνητική συνέβεια στο περιβάλλον. Τώρα για την οδηγία πλαίσιο για τα νερά. Οι πιο πρόσφατε πληροφορίε που διαθέτουμε, από Μάρτιο και Απρίλιο δηλαδή, δείχνουν ότι η Συνομοσπονδία για την χρήση των υδάτων του ποταμού Γουαδαλκιβίρ διαθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι θα υπάρχει αρνητική επίπτωση από τις αντλήσεις, υγειοτρήσεις μάλλον που έχουν εγκριθεί για τα νερά του ποταμού. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει ξεκάθαρα διαπίστωση αιτιόδου συνάφειας ανάμεσα στην άντληση υδάτων από τις γεωτρήσεις αυτές και στα επίπεδα του νερού στις διάφορες πηγές. Δεν γνωρίζουμε με άλλα λόγια αν έχει όντως συμβεί αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η οικολογική κατάσταση της λεκάνης αυτής εκτιμάται, καθώς επίσης και τα απαραίτητα να ληφθούν μέτρα, μέσα στα, μέσα στα πλαίσια του διαχειριστικού σχεδίου. Υπάρχουν και άλλα σχέδια τα οποία δεν διαθέτουμε, 23 συνολικά. Γι' αυτό η Κομισιόν απεφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Η γραπτή διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου έχει τώρα ολοκληρωθεί και αναμένουμε την έκδοση αποφάσεως. Περαιώνοντας, έχω να πω ότι η προκαταρκτική έρευνα δεν μας επέτρεψε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο παραβιάσεως και γι' αυτό η Κομισιόν αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία επί παραβιάση των τριών οδηγιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρυσι, στο τέλος του έτους, ήρθα στην Επιτροπή για να υποστηρίξω την αναφορά που κατέθεσε η πλατφόρμα για την ε, υπεράσπιση των πράσινων κοιλάδων και είχα μια ξεκάθαρη στάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι η υιοθέτηση των μέτρων που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος στην Ανδαλουσία και ειδικότερα στην περιοχή του Καδαλκιβίρ ε, με ανάκληση των αδειών που είχαν αποδοθεί και ε, δημιούργησαν τόση ζημιά στο πάρκο Σεγκούρα Ιλας ήταν αυτά τα θέματα τα οποία σας παρουσίασα. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω ε, και να σας καταθέσω και πάλι στοιχεία συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης του Διευθυντή του Φυσικού Πάρκου που ε, κάνει ξεκάθαρο το πρόβλημα. Ε, οι αρχές αποφάσισαν να περάσουν την έκθεση τους στις αρχές ε, που, που ασχολούνται με την ίδρυυση και το νερό στο Κουαταλκιβίρ. Γιατί <clears throat> στην έκθεση αυτή ε, αναφέρεται ότι δημιουργείται, ε, προκαλείται μάλλον ζημιά ανεπανόρθωτη στο, στην περιοχή του Κουαταλκιβίρ και στο φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται λοιπόν για μια τεχνική έκθεση του Διευθυντή του Φυσικού ε, Πάρκου. Εξαιτία λοιπόν της σοβαρότητας ε, και του ε, όλου πλαισίου θα ζητήσω από το Κοινοβούλιο να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να ζητήσει από την Κομισιόν να μάθει κατά πόσο θα ήταν καλό να προχωρήσει η διαδικασία επί και είναι σημαντικό ε, να ληφθεί υπόψη αυτή η τεχνική έκθεση ε, για την περιβαλλοντική ζημιά που έχει προκληθεί και να είναι ε, ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες για το περιβάλλον και τα πτηνά. Επίσης, οι ισπανικές αρχές θα πρέπει να εμπλακούν και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και προετοιμασίας για να μπορέσουν να διορθώσουν τη ζημιά που έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν φτάνει ως εδώ ένας αναφέρον, για δεύτερη μάλιστα φορά, όπως και ο ίδιος το επεσήμανε, είχε έρθει εδώ πριν από 4,5 μήνες, όταν έρχεται λοιπόν εδώ να μας εκετεύσει, να μας παρακαλέσει να αναλάβουμε δράση, διότι τίποτε απολύτως δεν έγινε, αυτό κάτι σημαίνει. Το επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα με προσοχή όσα είπε ο ο καθηγητής που πήρε το λόγο όμως, όταν μιλάμε για μια αναφορά που καλύπτει μια τέτοια έκταση και παίρνει τέτοιες διαστάσεις, σωστό είναι ότι πρέπει να συνεχίζει κανείς την προσπάθεια. Εγώ έχω να σας θέσω μια ερώτηση. Εσείς πότε, ρωτήσατε, πότε ζητήσατε για πρώτη φορά από την Ισπανική κυβέρνηση να σας δώσει πληροφορίες, έχετε συγκεκριμένη ημερομηνία, πότε ήρθατε σε επαφή για πρώτη φορά με τις Ισπανικές αρχές, ε, με την σημερινή ή την προηγούμενη κυβέρνηση ήρθατε σε επαφή. Και έπειτα, Πρόεδρε, βάσει των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω πρέπει να αναλάβουμε δράση. Όχι μόνο για να μην είναι ανοιχτή αυτή η αναφορά, αλλά για να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε και μία λύση. Μην ξανάρθει εδώ αναφέρω να μας παρακαλέσει, να λάβει πολύ γρήγορα δράση η Επιτροπή Αναφορών μας. Ευχαριστώ, κύριος Γιάρ. Κυρία Πρόεδρε, η ερώτησή μου είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση ε, με την παράκληση του συναδέλφου Ετελγκάης, αλλά να συμπληρώσω ε, επιπλέον ε, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί ως άμεσο ε, μέτρο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε περαιτέρω ζημιά. Ζητώ από την Κομισιόν, η οποία έχει αναφέρει σημαντικές αμφιβολίες ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή ενομοθεσία ε, να πω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία έχει κάποια διάρκεια ταυτόχρονα. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ε, αναστρέψουν αυτή τη βλάβη στο περιβάλλον. Αυτό που δεν μπορούμε να ανεχθούμε είναι να μαλώνουμε δύο-τρία χρόνια και τελικά όταν θα αποδειχθεί ότι έχουμε δίκιο ε, να έχει ε, το περιβάλλον υποστεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την τωρινή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και να ληφθούν άμεσα μέτρα. Να ζητήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποφευχθούν περαιτέρω ε, ζημιές, περαιτέρω βλάβες στο περιβάλλον. Να μην ε, μαλώνουμε λοιπόν τελικά για χρόνια και τελικά όταν αποδειχθεί ότι έχουμε δίκιο να μην υπάρχει πια αυτή η περιοχή φυσικού κάλους. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω πλήρωσε την πρότασή σας για ε, διερεύνηση δυνατοτήτων διαλόγου με την ε, κυβέρνηση ε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ευχαριστώ. Well, I'm, I'm confused. κυρία Λόικεν, ευχαριστώ, αλλά έχω περιέλθει σε σύγχυση. Ίσως να μην κατάλαβα καλά τη μετάφραση. Ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέντησε πολύ διαφορετικά από αυτά που είχα απέντησει στη γραπτή ε, απάντησή τους. Εξ όσων κατάλαβα, η Επιτροπή λέει ότι έχει μελετήσει το θέμα και ότι θα πρέπει να υπάρξει λύση από το δικαστήριο. Πήγε στο δικαστήριο λοιπόν, ενώ οι Ισπανοί μας λένε ότι συνεχίζει να μην γίνεται τίποτα. Μα, δεν άκουσα καλά. Μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προσέφηκε σε δικαστήριο ή όχι. Διότι ε, διαφορετικά θα πρέπει να είμαστε πολύ θυμωμένοι. Διότι διαβάζοντα τη γραπτή απάντηση, σκέφτηκα ότι πάμε από αναβολή σε αναβολή. Δεν γίνεται τίποτα και είμαστε συνεχώ στο μηδέν. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ακούσαμε μια νέα απάντηση. Μήπως παρανόησα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εάν μπορούμε, βεβαίω και να γίνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ και να καταλάβω τι θα είναι αυτό. Εάν μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση, η Ισπανική κυβέρνηση είναι που θα πρέπει να αναλάβει ευθύνε και να πάυσε την κατάσταση, εφόσον μιλάμε για δικαστική υπόθεση. Τι μας είπε ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, τι θέλουμε να κάνει για μας. Ο κύριος Μποσενάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή Επιτροπή, ίσως κάποια από εσάς να διαβάσατε το βιβλίο του Λέστερ Μπράουν, Plan B. Στο βιβλίο αυτό, ο κύριος Μπράουν περιγράφει μια υπόθεση σχεδόν πανομοιότυπη. μια περίπτωση που μοιάζει πολύ με το ποτάμο Γουαδαλκιβίρ στη Σαουδική Αραβία. Στα τέλη της δεκαετία του 1990 η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να αρχίσει ένα εντυπωσιακό εγχείρημα άρδευση χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ε, υδροφόρους ορίζοντες σε μεγάλο βάθος. Αυτό όμως οδήγησε σε σχεδόν ε, πλήρη εξάντληση των ε, υδροφόρων αυτών οριζόντων. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο σκληρή, ακόμη πιο οξία απερίμωση στην Σαουδική Αραβία η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί πια να αρδεύσει καθόλου καλλιέργειε. και εδώ, σε περιφερειακό ή κυβερνητικό επίπεδο, θα πρέπει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν αυτά που καταγγέλει ο κύριος Μπράουν είναι ορθά για το ευρωπαϊκό έδαφος δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί δεν κοιτάζεται εάν υπάρχει σωστή υλοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους υδροφόρους ορίζοντες. Είναι σαφή, σαφή όσα λέει η οδηγία αυτή για μένα. Αποξήρανση σημαίνει διαδικασία απερίμωσης. Αυτή η αποξήρανση των υδροφόρων οριζόντων σημαίνει ακριβώς εξαφάνιση της βιοποικιλότητας που επιδιώκουμε με το Natura 2000 λόγου χάρη. Πώς γίνεται να σπαταλάμε τόσο χρόνο παρακαλώντας τις ε, επιμέρους κυβερνήσεις ή τις κεντρικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει εάν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία στον ίδιο ρυθμό. Πρέπει να πάυσουν όλα αυτά, όχι μόνο στην περίπτωση της Ισπανίας. Είναι πολύ σημαντικό και επίγον να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ευθέτω χρόνο και να μην περιμένει και να περνάει ο καιρός. Οι πληροφορίες που λάβαμε σήμερα είναι ελλειπείς, δεν είναι επαρκείς και για να μην πω είναι και άστοχες. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποφάσισε να κοιτάξει τουλάχιστον τις δύο πτυχές την ορθή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τι ε, δυσμενείς συνέπειε, διότι δεν μιλάμε εδώ μόνο για υδροφόρου ορίζοντες που πλήττονται, αλλά και για αντίκτυπο τη αποξήρανση ε, και τη απερίμωση που πλήττουν τη βιοπικιλότητα στα πλαίσια του Natura 2000. Δεν είναι τόσο περίπλοκο να το κατανοήσετε και να υπάρξει κάποια αντίδραση. Ας διαβάζουμε ξανά και ξανά τα έργα του κυρίου Μπράουν και άλλων συγγραφέων. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά οι συνέπειες εντωμεταξύ είναι καταστρεπτικές. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και να αντιδράσουμε, αντί απλώς να καθόμαστε να περιμένουμε. Η αναφορά προφανώς να παραμένει ανοιχτή. Και να ζητήσουμε από την Ισπανική κυβέρνηση πληρέστατη, διεξοδική απάντηση για το πώς έχει κατάσταση. Να δούμε κατά πόσον ε, οι μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου έγιναν και διεξήθησαν με σωστό τρόπο και κατά πόσον η υλοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τους εντροφόρους ορίζοντες εφαρμόστηκαν σωστά. Εάν ελήφθησαν υπόψη οι δυσμενείς συνέπειες. Ιδάλλως θα πρέπει να αναλυφθεί δράση. Να πάψουμε να χάνουμε χρόνο. Ευχαριστούμε κύριε Μποσουνάρου. Κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να επαναλάβω τις ανησυχίες που ήδη έχουν ε, εκφραστεί. Καταρχάς, ε, θα προσπαθήσω να ε, καταλάβω τι ακριβώς μας λέει σήμερα η Κομισιόν εδώ και μας παρουσιάζει γραπτός και προφορικάς. και εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες όταν ε, κοιτάζω το έγγραφο που έχω εδώ, ε, την ανακοίνωση στα μέλη. Στο τέλος λέει ότι η Επίτροπη δεν μπορεί να, ε, να δώσει οποιαδήποτε συνέχεια στο θέμα του αιτήματο. Αυτό αναφέρεται στα στοιχεία της 26ης Ιανουαρίου. Αυτό που μας είπε προφορικά η Κομισιόν τώρα Ε, είναι, ε, έχει να κάνει με την διαδικασία επί παραβίαση. Ε, τι γίνεται τελικά, κάνει κάτι ήδη η Κομισιόν ή δεν μπορεί να κάνει κάτι περαιτέρω. Ποια είναι ακριβώς η στάση της Κομισιόν σήμερα, τι κάνει σχετικά με το θέμα, δεν κάνει τίποτα. Δεύτερον, Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ε, θέμα και σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά ε, και οικονομίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως και εδώ υπάρχει κάποια αντίστα, αντίφαση στα όσα διαβάζουμε. Ε, Natura 2000. Πλήρης παραβίαση της οδηγίας για το ε, οικοσύστημα. Βιότοπο. Κάπως προσπαθήσαμε να επιλύσουμε θετικά αυτή την αντίφαση με αυτή την ε, ε, ε, προσπάθεια να βρούμε μια επίγουσα λύση. Ε, αυτή η βιασύνη δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έλαβε ε, τα κατάλληλα μέτρα, αλλά με το γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα στην Ισπανία, από τις Ισπανικές αρχές. Αν δεν ε, προχωρήσει, παρόλο και αν δεν προχωρήσει εδώ η διαδικασία, χρειαζόμαστε μια γρήγορη λύση. Ευχαριστώ, συνάδελφος Άουγκεν. Ε, ευχαριστώ. Παρακολούθησα όσα είπε, όπως είπαν οι συνάδελφοι, αλλά εκπλήσωμαι. Εγώ αναγκαστικά ακούω τη διερμηνία. Φαίνεται ότι όσοι ακούν ε, ισπανικά κάτι άλλο καταλαβαίνουν. Όσοι λοιπόν ακούν άλλες γλώσσες όπως και εγώ, κατάλαβαν ότι και εγώ κατάλαβαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάση και παραμένει ένα ερώτημα για ένα σκέλος μιας οδηγίας και το κατά πόσο αυτό παρακολουθείτε. Με συγχωρείτε, εγώ νομίζω ότι η αναφορά αυτή πρέπει να κλείσει. Έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό η διαδικασία. Θα πρέπει να αποστείλουμε επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση προκειμένου να επιταχύνει και να μην περιμένουμε την εκδίκαση από το δικαστήριο. Είναι σοβαρά τα προβλήματα, εντάξει αλλά καμιά φορά κερδίζουμε και δεν θα πρέπει να υιοθετούμε τη στάση του ηττημένου. Έχει πάει καλά η όλη υπόθεση. Φαίνεται ότι είχαμε επιτυχία. Απλώ να καλέσουμε την Ισπανική κυβέρνηση να επιταχύνει τι διαδικασίε. Αυτή είναι η δική μου σύσταση. Θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Επιτροπή να αποσαφηνίσει την αμφιβολία που τελικά έχει δημιουργηθεί στον όλων των συναδέλφων. Υπέρξε μετεβολή στη στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη γραπτή απάντηση που μα απέστειλε και το τι μα λέει σήμερα. Διότι σε αυτή την περίπτωση είναι θετική η εξέλιξη. Όμω η εμφιβολία κάποιων συναδέλφων είναι σημαντική. Πού βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έχει εκκινηθεί διαδικασία, υπάρχει προσφυγή στο δικαστήριο ή όχι. Μπορείτε να μας το πείτε για να μπορέσουμε κι εμείς να αναλάβουμε λόγος δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω. Εάν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με τη διευκρίνηση αυτή που ζητήσατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε για τρίτη φορά στην Ισπανική κυβέρνηση και με ρωτήσατε σε ποια ημερομηνία. Τέλη Νοεμβρίου 2011. Η η Ισπανική κυβέρνηση απήντησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Ιανουαρίου 2012. Δεύτερον, ναι, υπήρξε μεταβολή στη στάση της Επιτροπής, σημαντική μάλιστα. Και σε σχέση με την προηγούμενη γραπτή μας απάντηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι στο μεταξύ μεταξύ της τελευταίας γραπτής απάντησης που αποστήλαμε στο Ευρωκοινοβούλιο και της σημερινής ημερομηνία έλαβε ουσιώδης πληροφορίες η Εκτελεστική Επιτροπή που ε, της ε, απέστειλε ο αναφέρον εκεί. Αποδεικνύεται ότι οι αρχές διαχείρισης αυτού του χώρου διαπιστώνουν σχέση αιτίωτη ατού μεταξύ της εξόρυξης υδάτων και των συνεπειών που έχουν υποστεί όχι μόνο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και τα οικοσυστήματα αυτής της περιοχής. Επίσης, η ανάλογη οδηγία ε, επιβάλλει τη δειγματοληψία ε, στο έδαφος της περιοχής. Απλώς σήμερα δεν μπορούμε ακόμη να αποκλείσουμε την υπόθεση να έχει πληγεί το φυσικό τοπίο της περιοχής ακριβώς λόγω αυτής της διαδικασίας. η εξόριξη τος η άντληση υδατός από τους υδροφόρους ορίζοντες μπορεί λοιπόν να έχει σοβαρά, σοβαρές συνέπειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας ε, για τα ύδατα, για τους υδροφόρους ορίζοντες και τις υδάτινες λεκάνες, εκεί Όντω δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Γι' αυτό απευθύνθηκε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, εφόσον μιλάμε για αρχές της οικολογίας, για υδάτινα αποθέματα που πρέπει να προστατεύονται μέσω των υδροφόρων οριζόντων, όλα αυτά θα μας αποσχολήσουν ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που παραβάσει. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσον υπάρχει παράβαση ως προς τις οδηγίες για την προστασία των οικοτόπων και για τα ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα φροντίσει να προχωρήσει όλη τη δικασία. Η όλη διαδικασία παραβάση θα συζητηθεί και στο σώμα των επιτρόπων. Απλώ δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά μόλι έχουμε περισσότερα στοιχεία, θα σα ενημερώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε το θέμα όσο το δυνατόν ε, πιο άμεσα. Κυρίω Στρουγκάη. Ευχαριστώ. Η δική μου ερώτηση ε, δεν απαντήθηκε ακριβώς. Αυτό που είπε η Κομισιόν ήταν ξεκάθαρο. Είπε ότι έχει καταθέσει έτοιμα στις Ισπανικές Αρχές τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Ε, τώρα όμως, ε, ε, εφόσον έχει, αλλαγή, έχει υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης, πρέπει να ενημερώσουμε τη νέα κυβέρνηση σχετικά με το τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για διαδικασία επί παραβάση. Ε, ο Διευθυντής Ιδάτων της Νέας Ισπανικής ε, Κυβέρνησης πρέπει να ε, γνωρίζει ξεκάθαρα τι συμβαίνει με αυτή την αναφορά. Να γνωρίζει ότι σύρεται εδώ και μήνες αυτή η αναφορά και θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει μια ξεκάθαρη λύση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το βήμα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να είμαστε δηλαδή απολύτω ξεκάθαροι σχετικά με το που βρισκόμαστε δεδομένου του νέου κλίματος, δηλαδή της νέας κυβέρνησης στην Ισπανία. Τώρα, η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, δεν ξέρω αν το βάλαν σε κάποιο σιρτάρι, αλλά πρέπει να δώσουμε στη νέα κυβέρνηση τη δυνατότητα να μάθει περισσότερα για αυτό το θέμα, ε, ώστε ο νέος ε, υπεύθυνο της κυβέρνησης για αυτό το θέμα να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ε, στην Επιτροπή μας. Ο συνάδελφος Γκάρσης. Ευχαριστώ. Μόνο ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Ιτορκάης. Ακούσαμε να λέει ε, ο, το εκπρόσωπο της Κομισιόν να λέει ότι ε, τον Ιανουάριο δόθηκε η απάντηση και τότε ήδη υπήρχε η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα λόγω στον αναφέροντα για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή ε, ιδιότι κάνει πολύ καλή δουλειά με λίγα μέσα. Ξέρω ότι η δουλειά σας αξίζει το σεβασμό μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που μίλησαν και κατανόησαν την ουσία και το επίγον του ζητήματος. Πολύ σύντομα, να πω αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο φαίνεται ότι ε, σύμφωνα με την Κομισιόν φαίνεται ότι υπάρχουν ε, εύλογες αμφιβολίες. Ε, φαίνεται, ίσως, υπάρχει δηλαδή μια σειρά θεμάτων εδώ που ενδεχομένω ίσως φαίνεται να, ότι πρέπει να αποδειχθούν και τώρα η αρμόδια αρχή πρέπει να κάνει ε, μια έρευνα. Ε, εντάξει, από νομική άποψη το κατανοώ και ίσως αυτό ε, πρέπει να γίνει. Όμως, ως Ευρωπαίος πολίτης θα έλεγα ότι εδώ ε, δημιουργείται ανεπανόρθωτη ζημιά, το είπα στην αρχή και το επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πάρουμε επίγοντα μέτρα, χρειάζονται άμεσα μέτρα. Και αυτό ε, μπορεί να σημαίνει και αναστολή της άδειας. Όσο διεξάγονται οι έρευνες, όσο αναλύονται τα στοιχεία. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι ε, λόγω ε, ξεκάθαρα νομικών ζητημάτων να έχουμε τελικά, να καταλήξουμε τελικά με τελείως ανεπανόρθωτη ζημιά. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνική ευθύνη, όπως είπατε. Η Ισπανική κυβέρνηση πρέπει να λάβει και αυτή την πτυχή υπόψη της όταν αναλαμβάνει μέτρα. Είναι επίσης αλήθεια ότι δεν μπορούμε να εναντιονόμαστε στα συμφέροντα ε, ε, κάποιων πολιτών έναντι ε, συμφερόντων 350 εκατομμυρίων ε, πολιτών ε, που θίγονται από τα θέματα της Natura 2000 πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα δικά τους λοιπόν συμφέροντα. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και να συμφωνήσω με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την ανάγκη ενημέρωση ε, της ε, τρέχουσας κυβέρνησης για το τι συνέβη ε, στο παρελθόν. Ίσως οι αποφάσει να μην ήταν οι κατάλληλε, αλλά τώρα είναι στο χέρι της να τι διορθώσει. Σύντομα, επίσης, να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς που μας υποστηρίζουν σήμερα στις προσπάθειές μας και οι διερμηνείς σα ευχαριστούν. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε με την πρόταση αυτή να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά να προωθήσουμε έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήδη σημείωσε ότι έχει πραγματοποιήσει βήματα πρόοδου ώστε να επιταχυνθεί η επιπαραβάση διαδικασία. Ενδεχομένως να απευθυνθούμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ζητήσουμε αμέσως να ανακληθούν οι άδειες για το έργο. Διότι οι ανησυχίες που ακούστηκαν μέσω των παρεμβάσεων που ακούσαμε σήμερα θα πρέπει να καλυφθούν με την πρόληψη πρώτα απ' όλα της ζημίας και μετά με ενδεχόμενη ανάκτηση της αποκατάσταση της κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν ως κοινοβούλιο όχι να πολιορκήσουμε ακριβώς την περιφερειακή κυβέρνηση μόνον, αλλά να δώσουμε πράσινο φως και στις δύο διαδικασίες αυτές ταυτόχρονα. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, να κλείσουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό με αυτήν ακριβώς την απόφαση. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Υπαριθμών 6. Αναφορά Πορτογάλου πολίτη, εξ ονόματος της Πορτογαλικής Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΑΕΤΠ σχετικά με λυπή διαφάνεια στο πλαίσιο αιτήσεων ενίσχυσης από τα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρίσταται ο κύριος Ντεμάτος, εξ ονόματος των αναφερόντων. Του δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω την οργάνωση αυτή τη δεύτερη συζήτηση τη αναφορά που υποβάλαμε τον Ιούλιο του 2009 στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα να χαιρετήσω και του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλου του υπευθύνου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Η αναφορά μα γύρει ζητήματα οικονομικά και κοινοτικού δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ω νέο επιχειρηματία και σε αυτή την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχω αισθανθεί μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκεια σε σχέση με την καθυστέρηση των ευρωπαϊκών φορέων ώστε να αποφανθούν για το κατά πόσον είναι σωστή η στάση του κράτους μας για την προώθηση των ε, επιχειρηματικών πρωτοβουλειών στην Πορτογαλία. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα όσο και αν έχει γίνει ευάλωτο λόγω της κακής κατανόησης των Ευρωπαίων ηγετών. Η νεαρή μας ένωση υπέβαλε την ε, αναφορά αυτή τον Ιούλιο του 2009, επισημένοντας παραβιάσεις, καταχρήσεις και παρανομίες από την πλευρά του κράτους, οι οποίες παραβιάζουν βασικούς κανόνες της αγοράς και του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Πλήτεται η υγιής και ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πορτογαλίας. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα μετά την ε, συζήτηση τη αναφορά της 25 Ιανουαρίου 2011 που δεν έδωσε αποτελέσματα, να φύγουμε με σαφή εικόνα για το κατά πόσον είναι νόμιμη ή παράνομη αυτή η επιβάρυνση και η επίσημη κατοχή από το κράτος των επιχειρηματικών ε, δράσεων πρόθεση βάσει του νομοθετικού διατάγματος 191-2009 τη 17 Αυγούστου. Εδώ λοιπόν θα θέλαμε μια επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν έχουμε λάβει από το Σεπτέμβριο του 2009 και ε, διερεύνηση από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ζητηθεί από τα τέλη του 2009. Ε, σήμερα θέλουμε ακριβώς κάποια οριστικά συμπεράσματα για το κατά πόσον και ποιο είναι υπεύθυνο για το μοντέλο ανταγωνισμού που θα επιτρέψει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προώθηση από επιχειρήσεις στην Πορτοκαλία και στον Ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα. Νομίζουμε ότι οι τεχνικοί οργανισμοί του ΚΡΕΝ για την θεσμική προώθηση και την επιχειρηματική προώθηση έχουν οδηγήσει σε μια περίεργη σύγχυση. Είναι λοιπόν σημαντικό οι δράσεις της, ε, Ευρωπαϊκής, της κυβέρνηση και του Πορτογαλικού ε, κράτου από το 2009, τον Αύγουστο του 2009, να εξεταστούν προσεκτικά, διότι υπάρχει ακριβώ συγχώνευση με τις ε, επιχειρηματικέ δράσεις προώθησης. Εδώ μιλάμε για προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών του τουρισμού, αλλά και για ε, επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις εμπορικού χαρακτήρα με υπηρεσίες και δράσεις που ε, με εκστατείες προώθησης μπορεί να έχουν οικονομική στήριξη. Αυτή η παράνομη, παραβατική, κρατική στάσεις στον τομέα των, επιχειρηματικών, των δράσεων προώθησης από τις επιχειρήσεις στην Πορτογαλία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, ιδίως με υποψηφιότητες επιχειρήσεων για το σύστημα στήριξης ε, που υπάρχει στην ε, χώρα και στον τομέα του τουρισμού. Εδώ λοιπόν να ότι στο εδάφιο ε, σίγμα του σχετικού κώδικα της Πορτογαλίας ανατίθεται στο, πορτογαλικό κράτος σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο να διασφαλίσουν την εύρωστη λειτουργία των αγορών, να υπάρχει ισόρροπος ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και να μην υπάρχουν παραβιάσεις μεταξύ μονοπωλιακών και καταχρηστικών δεσποζουσών θέσεων. Εδώ λοιπόν, εφόσον η αναφορά μας ήδη από τον Ήλιο του 2009 εξετάστηκε για πρώτη φορά, έχουν προθεθεί τρει ή τέσσερι ε, προπολογισμοί του κράτους, χωρίς, με μάλλον κοινοτικά κονδύλια να στηρίζουν τον τουρισμό, αλλά χωρίς να έχει αποσαφινιστεί αυτό το θέμα των παράνομων και κατακριστικών δράσεων, της ε, κρατικής παρέμβασης στον τομέα της τουριστικής ε, ε, προώθησης στην Πορτογαλία. Ήδη το 2009 έχουμε καταγγείλει αυτήν την ε, παράνομη παρέμβαση, ακόμα και στην ε, Βουλή Τη Πορτογαλική Δημοκρατία, όπου επισημάνθηκε από βουλευτέ διαφόρων κομμάτων ε, το τι κάνει η κυβέρνηση τη Πορτο... της για το πραγματικό αυτό πρόβλημα που δημιουργεί ένα μονοπόλιο και αρνητική ε, συμφόρηση τη ελεύθερη επιχειρηματική ε, τουριστική δραστηριότητα στην Πορτογαλία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε και στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και στους ηθήνοντες ώστε να γίνει πραγματικά κάτι για την κατάσταση αυτή. Η νεαρή μας ε, οργάνωση ε, θα πρέπει να απευθυνθεί, μάθαμε και σε ανώτερα δικαστήρια, ώστε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Λισαβόνας να ε, εξεταστεί για δεύτερη φορά. Εκεί επισημάνθηκε, ελήφθη απόφαση μάλλον, σε σχέση με την επικάλυψη κοινών προγραμμάτων και των όσων προβλέπονται για τους συγκεκριμένους, για τους υπεύθυνους οργανισμούς του Κρέν, κάτι που σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα σαν το δικό μας θα απορριφθεί. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Επιτροπή σας θα καταλάβει την σημασία που θα έχει η στάση της στο να παρεμποδιστεί αυτή η αρνητική προσπάθεια της κρατικής παρέμβασης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες πρόθεσης στην Πορτογαλία. Και βεβαίως ανάλογα με και με την οικονομική ε, κατηγοριοποίηση της νίκαιας ε, στην τάξη 35. Εδώ λοιπόν στην Πορτογαλία θέλω να πω ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και από κοινωνική και οικονομική άποψη το ελεύθερο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Για άλλη μια φορά, να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα και την ευκαιρία που μα δώσατε σήμερα να παρουσιάσουμε την αναφορά μα. Ευχαριστώ όλου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής χαιρετώντας και τους υπευθύνους της Πορτογαλικής Αντιπροσωπείας που παρέστονται στην αίθουσα Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε εγώ θα μιλήσω εκπροσωπώντας την Γενική Διεύθυνση Ρέτζη και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αν συμφωνείτε. Πολύ καλά, είστε ο κύριος Καρντόζο, λέει. Δηλαδή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα να δώσω κάποια στοιχεία σε σχέση με την αναφορά αυτή. Όπως παρουσιάστηκε η αναφορά αυτή στην Επιτροπή Αναφορών ήδη εδώ και ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2011. απλώς εγώ να θυμίσω κάποια πράγματα που υπόθηκαν πριν από ένα χρόνο. Να θυμίσουμε το γενικότερο οποίο μια αναφορά που είναι παλιά, χρονολογείται από το 2009. Αφορά πρόγραμμα που έβαλε ο αναφέρον για ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια στα πλαίσια της πολιτικής ε, συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών ενημέρωσαν τον αναφέροντα ότι βάσει του συστήματος επιλεξιμότητας των προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία, η αρμοδιότητα για την εξέταση, την επιλογή και την τελική χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανήκει στα κάτι μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητες νομικέ αρμοδιότητε για να διαχειριστεί απευθεία τέτοιου είδου προγράμματα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζουμε ότι έγινε στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι να επαληθεύει εάν σε γενικέ γραμμέ υπήρξε παραβίαση των όσων προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό νομίζω το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή σας ε, στις αρχές Ιανουαρίου 2011 ενημερώθηκε σχετικά και από τη μια σε ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο στην Πορτογαλία η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν ε, υπήρξε παραβίαση. Ε, ενημερώσαμε σχετικά και τον αναφέροντα και θεωρήσαμε ότι έκλεισε υπόθεση. Δεν υπήρξε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Τώρα, προ τα κριτήρια επιλεξιμότητα και χρηματοδότηση ε, των προγραμμάτων, ενημερώσαμε τον αναφέροντα και την Επιτροπή σα ότι οι διαδικασίε ε, υλοποίηση είναι εθνικού χαρακτήρα. Τα αρμόδια δικαστήρια για να λάβουν και να εξετάσουν τέτοιες προσφυγές για την ε, έγκριση απόρριψη προγραμμάτων είναι ακριβώ τα εθνικά δικαστήρια τα, τα στοιχεία αυτά τα αποστήλαμε και στον αναφέροντα. Τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας του ακριβώς εξετάζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τέλος, ένα τρίτο σημείο, γενικές σκέψεις για τους μηχανισμούς μάλλον τους ε, μηχανισμούς, την αξιολόγηση των μηχανισμών αποτίμησης. Εμείς κάναμε μια τέτοια αξιολόγηση στην Πορτογαλία και ω προς τη διαφάνεια των μηχανισμών τις λεπτομερείς που θα πρέπει να αποστέλλονται στου ε, υποψηφίους, τους υποβάλλονται στα προγράμματα. Είδαμε τι προσπάθεια έγινε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να λάβουμε πληροφορίες από την Πορτογαλία, αλλά δεν μπορέσαμε να επηρεάσουμε τις τελικές αποφάσεις για την ανάθεση όχι ε, προγραμμάτων. Εδώ βεβαίω πάλι μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση σε εθνικό επίπεδο, εφόσον απευθυνθεί κανεί, αποταθεί στα εθνικά δικαστήρια. Τώρα, σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το 2011 ήδη είπαμε στην ε, Επιτροπή σα ότι θεωρεί λίκασα την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω, περαιτέρω εξέταση τη ε, αναφορά θα πρέπει να υπάρξει ιδίω ω προ την ε, σύλληψη και την παροχή τη κρατική επιδότηση. Τώρα για το κατά πόσο υπήρξαν εξελίξει από τον Ιανουάριο του 2011 να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τη Γενική Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ω προ το θέμα αυτό... Η, η Κομισιόν ζήτησε από του αναφερομένους περισσότερε πληροφορίε για τι κρατικέ επιδοτήσει σχετικά με την αρχική αναφορά και τι λάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2011 προχωρήσαμε σε αλληλογραφία με τις ε, πορτογαλικές αρχές από τότε. Το θέμα των κρατικών ενισχύσεων τίθεται εκεί όπου η δημόσια αρχή χορηγεί δημόσια χρήματα ενώ, ε, ε, για ενίσχυση δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν οι ίδιες ανάγκες να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι το παράπονο. Αυτή είναι η καταγγελία δηλαδή των αναφερομένων. Τώρα, το πορτογαλικό, η πορτογαλική υπηρεσία τουρισμού μας απήντησαν δεν ασκεί τέτοιες δραστηριότητες. Εμείς αναμένουμε και άλλες πληροφορίες και θα δώσουμε απάντηση σήμερα την επεξεργαζόμαστε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στον αναφερόμενο μέχρι το Σαββατοκύριακο. Με συγχωρείτε, Μέχρι τι διακοπέ. Ευχαριστούμε. Δεν φαίνεται να υπάρχουν όμω άλλε παρεμβάσει, οπότε να ακούσουμε τον αναφέροντα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι, της... υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας εξήγησαν τις απόψεις τους, όμως υπάρχει ένα θέμα, να το πω αυτό στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζη, σε σχέση με την εθνική νομοθεσία, σε σχέση με τις προσπάθειές μας, φαίνεται ότι de facto υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων σε κρατικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα εξέταση της υπόθεσης δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κλείσιμο της υπόθεσης χωρίς να υπάρχει οριστική εξέλιξη. Να πω λοιπόν στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεθνής ότι αν για κάποιο λόγο, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίσει ότι το νομοθετικό διάταγμα 2001, μάλλον 191 το 2009, παραβαίνει τους κανόνες ανταγωνισμού. Κάτι που εμείς το επισημαίνουμε στην Πορτογαλία επανειλημμένος σε, σε, σε επίπεδο Συμβουλή Επικρατείας. Εδώ δεν θα θέσει ένα αμφιβόλο η όλη στάση της Πορτογαλίας στη συγκεκριμένη υπόθεση την ανάπτυξη του περιφερειακού ανταγωνισμού. Διότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι δεν καταλάβαμε τι αφορά η υπόθεση. Οι τεχνικοί οργανισμοί του ΚΡΕΜ που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση αναγνώρισαν ενώπιον δικαστηρίου με αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν εκεί ότι έχουν ουσιαστικά ε, απορρίψει την ε, υποψηφιότητά μας διότι δεν υπήρξε συμφωνία, δεν υπήρξε συντονισμός με τους στόχους του όλου προγράμματος. Μα ε, μπορεί ένα τεχνικό οργανισμό που έχει εμπορικέ φιλοδοξίε ε, σε ένα συγκεκριμένο ε, τομέα να κρίνει ένα άλλο οργανισμό ή μια ένωση που έχει επίση εμπορικέ φιλοδοξίε στον ίδιο τομέα, εγώ το αμφισβητώ αυτό. Διότι προφανώ το αποτέλεσμα για μένα είναι λογικά προφανέ και θα πρέπει να ε, αγωνιστούμε και στα δικαστήρια. Έχουμε να κάνουμε με κρατική επίθεση εδώ. Κατά εμπορικής δραστηριότητας που το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένε υποχρεώσει να αποσαφηνίσει την κατάσταση αυτή. Τα ευρωπαϊκά ταμεία που ε, αναλογούν στην Πορτογαλία, πρέ, ε, αναλογούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων της Πορτογαλίας ή μόνο για κρατικούς φορείς που βλάπτουν, ζημιώνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ε, που δεν ανήκουν στο κράτο. Θέλουμε αυτό να αποσαφινιστεί. Μιλάμε εδώ για μια πραγματική επίθεση. Για ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει. Αυτό δεν μπορούμε να το παραμερίσουμε. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και σε επίπεδο τη Ευρώπη ολόκληρη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Σα ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον σε σχέση με τα αιτήματα που έχουμε εκφράσει εξ ονόματος των αναφερόντων για δεύτερη φορά τους έχουμε μεταβιβάσει η απάντησή σας δεν είναι καλή πλήρης και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνεργασία αλλά για άλλη μια φορά θα ήθελα να κατακρίνω την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν μας επιτρέπει να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που εκφράζουν οι αναφορές των πολιτών. Θα φροντίσουμε λοιπόν να αποστείλουμε επιστολή στις πορτογαλικές αρχές καταγγέλλοντας και για δικό μας το λογαριασμό τα όσα συμβαίνουν. Θα απαιτήσουμε απαντήσεις. Νομίζω εντωμεταξύ έτοιμα πρέπει να απευθύνουμε και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να κατακρίνουμε ακριβώς, να επικρίνουμε την ε, συμπεριφορά τους, τη στάση τους. δεν αρνήθηκαν τι αρμοδιότητέ του ε, στι γραπτέ του απαντήσει τη σημερινέ του παρεμβάσει οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει αρμοδιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί και δράση και η ευθύνη αναλόγω. Ο εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζη ζητά και πάλι ο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να αντιδράσω στα όσα είπα αναφέρον. Να διευκρινίσω ότι εδώ δεν μπορούμε να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειε. Από το 2009 ω σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ συγκεκριμένα στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης έχει μια τεράστια αλληλογραφία για το θέμα αυτό. Έχω όλο αυτό το σχέδιο δίπλα μου και ευχαρίστως να σας δώσω τον τόμο με τις πληροφορίες και τα στοιχεία. Καθορίσαμε ότι η διαχείριση ε, των Ευρωπαϊκών Ταμείων Στήριξης, όπως το ΦΕΝΤΕΡ, είναι αρκετά περίπλοκη. Εδώ μιλάμε για προγράμματα που ξεπερνάνε τα 5.000. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά να τα διαχειριστεί μόνη τη. Και αυτό με πλήρη συνείδηση και έχοντα κατά την άποψή μα ρωτήσει και ζητήσει όλες τις απαραίτητε πληροφορίες από την ε, Πορτογαλική αρχή, από τις Πορτογαλικές αρχές. Εξετάζοντα και συλλέγοντα μάλλον και εξετάζοντα όλε αυτέ τι πληροφορίε, θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Αυτό που είπαμε στον αναφέροντα είναι ότι τα ζητήματα αυτά που εκκρεμούν, γιατί αναφερθήκατε για το συνταγματικό σας δίκαιο, είναι ζητήματα πρέπει να λυθούν σε εθνικό επίπεδο. Διοικητικά δικαστήρια, συνταγματικά δικαστήρια τη Πορτογαλία όμω. Δεν μπορεί να τα αναλάβει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μα ευθύνη αφορά το ερώτημα το κατά πόσον υπάρχει παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό το έχουμε αποστείλει στους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Το είπα αυτό και νομίζω ότι έχουμε πληρώσει την αποστολή μας. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ευχαριστώ και τους αναφέροντες. Ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση όσο το δυνατόν συντομότερα. Κλείνουμε με το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Γνωμοδότηση με θέμα πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια του συναδέλφου Βάλεαν. Σήμερα όμως δεν μπορούσε να παρίσταται. Η συνάδελφος Νικολάη έχει πάρει τη θέση του για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Δεν μπορεί δυστυχώς να είναι παρούσα η συνάδελφός μου σήμερα. Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε το πρόγραμμα για την Ιθαγένεια 2014-2020 τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερος αριθμός αναφορών καταχωρούνται σχετικά με την παρεμπόδιση πολιτών να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, 45% του αριθμού των αναφορών που λαμβάνουμε έχουν σχέση με το θέμα αυτό και σύμφωνα με τη Citizen Report του 2010 η συνηθέστερη καταγγελία είναι οι δυσκολίε λόγω των πρόσθετων γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων, οι καθυστερήσει από πλευρά τη διοικήσεω στην ε, ε, χορήγηση αδειών διαμονή και ούτω καθεξής. Τον Οκτώβριο του 2010 είχαμε 63 ε, περιπτώσεις παραβιάσεων που ήρθαν ενώπιον των δικαστήριων δηλαδή. Επίσης διαπιστώνουμε έλλειψη ενημερώσεως από πλευράς πολιτών σχετικά με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και ε, για τις συνθήκες, τη συνθήκη μάλλον, ε, δικαιωμάτων ανθρώπων με αναπηρίες. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις διατάξεις των δύο αυτών εγγράφων και γι' αυτό σημειώνονται και συχνές παρανοήσεις. Η προκείμενη υπόθεση Μάλλον για να αντιμετωπιστεί το θέμα, να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αυτή ενημέρωσης, γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης, κατάρτισης. Το πρόγραμμα του 2014-2020 που διαδέχεται το προηγούμενο πρόγραμμα, όπως γνωρίζετε, αναμένεται να δώσει απλούστερη μορφή και ορθολογικότερη μορφή με ταχύτερους στόχους και πιο καλή διαχείριση των πόρων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στο να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και να δοθούν οι προτεραιότητες με καλύτερο τρόπο. Δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απαραίτητη ευελιξία για να μπορέσει να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες που προκύπτουν. Ωστόσο, έχω ορισμένε ανησυχίε σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα γιατί η πρόβλεψη για το 2014, δηλαδή Ιανουάριο 2014 μέχρι Δεκέμβριο του 2020, όπως γνωρίζετε, είναι τη τάξη των 439 εκατομμυρίων, που βρίσκω ότι δεν είναι ρεαλιστικό το ποσό αυτό, διότι υπάρχουν και πρόσθετες πτυχές στο πρόγραμμα και τελειώνει το πρόγραμμα του 2007-2014 και αυτή, αυτή η έλλειψη θα, είναι, θα έχει αρνητικέ συνέπειε. Το νέο πρόγραμμα δεν πρέπει να καθυστερήσει και πρέπει να είναι επιχειρησιακό ευθύ εξ αρχή, από την αρχή του έτους 2014. Αυτές είναι οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. Σημειώνονται ακόμα σημαντικές ανισότητες, ιδίω θέματα βίας κατά των γυναικών εξακολουθούν να είναι η χειρότερη έκφανση αυτής της ανισότητας. Μία πτυχή του προγράμματος αναφέρεται στην καταπολέμηση της βίας και κυρίως της οικιακής βίας. Η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει σημαντικό αριθμό αναφορών που αναφέρονται στους στόχους του προγράμματος και ορισμένοι αναφερόμενοι αλλά και οργανώσεις σημειώνουν τη μεγάλη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης και κυρίως για τα εθνικά προγράμματα τα οποία υποβάλλονται από μικρές μη κρατικές οργανώσεις. Χρειάζεται διαφανής κατανομή των κονδυλίων όχι μόνο στα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και στις μικρότερες οργανώσεις. Υπενθυμίζω στις και στους συναδέλφους ότι η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 24 Μαΐου. Θα συζητηθούν οι τροπολογίες αυτές στις 19 έκτου. Η έγκριση της γνωμοδοτήσεως προβλέπεται να γίνει στις 12 Εβδόμου. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να εγκαταλείψω την αίθουσα γιατί πρέπει να προεδρεύσω αλλού. Κολέγα Μποσινάρου. Ο κύριος, Μποστινάρου. Μιλώ εξ ονόματος του κύριου Κάσμαν, του συναδέλφου μου, που είναι δυστυχώς ε, απόν σήμερα, ε, κολλείεται δηλαδή. Ευχαριστούμε την κυρία Βαλεάν για τα λόγια της, για το πρόγραμμα προστασίας των πολιτών για το 2014-2020. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επιτακτικό ναι μεν η Επιτροπή μας δίδει απλώς, γνωμοδότηση, αυτή όμως πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη. Είναι σημαντικό στη γνωμοδότησή μας να επιμείνουμε ώστε το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια 2014-2020 να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας. Η Επιτροπή μας πρέπει να διευρύνει τους στόχους του προγράμματος, να προσθέσει και νέους στόχους δηλαδή, έτσι ώστε να δοθεί το σωστό μήνυμα προς ε, τους πολίτες ότι δικό τους είναι το πρόγραμμα αυτό θα μελετήσουμε την υποβολή τροπολογιών στην ε, γνωμοδότηση και θα εξετάσουμε και ορισμένα θέματα κυρίως γλωσσικών διατυπώσεων και συνεκτικότητας. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Ο κύριος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η κυρία Σρέτερ θέλει να παρέμβει. Όχι. Να θυμίσω Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 24 Μαΐου, όπως τόνισε ο συνάδελφος Νικολάη. Οι τροπολογίες έπειτα θα εξεταστούν στις 19 Ιουνίου και ψηφοφορία στις 12 Ιουλίου. Οι σκέψεις που μας παρουσίασε η κυρία Νικολάη σήμερα, βάσει του εγγράφου της κυρίας Βάλεαν, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και όπω επεσήμανε και ο κ. Μποστινάρου, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε βεβαίω έτσι περαιτέρω το κείμενο, ώστε να δώσουμε και εμεί τη συνεισφορά μα. Κλείνουμε με το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο. Με γνωμοδότηση σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο τη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 2010. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γκέρινγκερ. Κυρία Γκέρινγκερ, συγγνώμη. Ε, Opinię, którą e, przygotowałam... E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση που ετοιμάσαμε βασίζεται στα στοιχεία και της έκθεσης της Ευρωπαϊκής της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Εδώ Μα απασχολεί το κατά πόσον έχουμε ορθή υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου και να εντοπίσουμε κενά και ελλείψεις. Η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Αναφορών, πρέπει να υπογραμμίσει κυρίως τις ελλείψεις κατά κενά. Ακριβώς διότι αφορά τη ροή προσφυγών και αναφορών που λαμβάνουμε στην Επιτροπή μας. Από τη δική μας τη Σκοπιά είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό. Οι πολίτες και οι ενώσεις πολιτών πολύ συχνά προσφεύγουν στο σύστημα των αναφορών για να εντοπίσουν περιπτώσεις μη σεβασμού του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη-μέλη. Προσπαθούν έτσι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να τα προστατεύσουν. Η Επιτροπή Αναφορών έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στην περίπτωση τέτοιων διεκδικήσεων τώρα στην... στον τομέα των αρμοδιοτήτων μας μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί ή ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις που αφορούν και ενδιαφέρουν περισσότερο τα δικαιώματα των πολιτών. Έχουν να κάνουν κυρίως με το περιβαλλοντικό δίκαιο και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και στο μέλλον. Ευτυχώς μπορούμε να πούμε ότι τα περισσότερα από τα, οι περισσότερες από τις αναφορές που λαμβάνουμε αφορούν ακριβώς αυτούς τους τομείς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να φροντίσει να υπάρξει καλύτερη υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη-μέλη και προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις σημαντικές καθυστερήσεις στην μεταφορά του κοινοτικού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Διότι αυτή ακριβώς εμποδίζει τους πολίτε να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους. Δικαιώματα τα οποία θεωρητικά έχουν γίνει αποδεκτά αλλά δεν εφαρμόζονται στις χώρες του. Μεγάλη σημασία έχει και το μεγάλο πιλωτικό πρόγραμμα που επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας αναφοράς του κάθε πολίτη. Ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν 18 χώρες μέλη. Ως τον Ιούλιο του 2010, 80% των υποθέσεων είχαν θεωρηθεί αποδεκτές και είχαν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει τη σημασία του πιλωτικού προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο κατά πόσον οι υποθέσεις αυτές ε, βρήκαν κάποια ευνοϊκή λύση ή όχι. Εγώ έχω εργαστεί επί δύο χρόνια στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και μπορώ να δω το θέμα αυτό και από τη σκοπιά της μιας Επιτροπής και της δικής μας. Ε, ανησυχία μας αφορά το γεγονός ότι οι αναφορές που απεστάλησαν στην Επιτροπή μας πολλές φορές αναπέμφθηκαν στα κράτη-μέλη προέλευσης του αναφέροντος και αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη κατάσταση ο πολίτης, ο αναφέρον τελικά βρέθηκε, βρισκόταν να πρέπει να λύσει το πρόβλημα που τον απασχολούσε στα πλαίσια του κράτους το οποίο κατήγγειλε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα, πιλωτικό πρόγραμμα, να το αποτιμήσουμε σωστά. Αρκετές είναι οι αναφορές που εξετάστηκαν, αλλά τελικά βρήκαν κάποια λύση ή όχι. Μήπως τελικά απορρίφθηκαν από το ίδιο το κράτος που καταγγελόταν. Δεν είναι πολύ λογικό να πρέπει κανείς να απαντήσει σε προσφυγή που στρέφεται εναντίον του. Θα πρέπει λοιπόν τα δικαιώματα των πολιτών να προστατεύονται επαρκέστερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης υπάρχει ανάγκη περισσότερης διαφάνειας και μεγαλύτερης επικοινωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου και για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα και για τους μελλοντικού μηχανισμούς που θα θελήσει να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές και τις παραβάσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε ορθότερη υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη-μέλη και βεβαίως την ε, γνώση από την πλευρά των πολιτών ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να θέλει να παρέμβει. Όχι. Υπογραμμίζω ότι και για την γνωμοδότηση αυτή προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στις 21 Μαΐου. Ψηφοφορία προβλέπεται στις 19 Ιουνίου. Την Επιτροπή Εκπροσωπείου Καλυφών Κέμπης Θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε εν συντομία την έκθεση και όχι απλώς να ε, απαντάμε στις παρατηρήσεις του εισηγητή. Ε, καταρχάς να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που Ανέφερε και τα θετικά σημεία, τις δυνατότητες που χρησιμοποίησε η Κομισιόν ε, πριν να ξεκινήσει τις πλήρες διαδικασίες ε, επιπαραβιάση. Το ποσοστό που αναφέρθηκε στην πρώτη έκθεση που κάναμε επιβεβαιώθηκε από μια πρόσφατη έκθεση την οποία θα έπρεπε να έχετε και την υιοθέτησε η Κομισιόν φέτος Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ε, το δεύτερο θετικό που αναφέρεται και στην έκθεση και σας ευχαριστούμε που το περιλάβατε είναι ότι οι παραβιάσεις είναι ένα κομμάτι στον κύκλο ζωής μιας νομοθεσίας. Ε, η λέξη κλειδί θα ήταν έξυπνοι, ε, έξυπνοι κανονισμοί. Όσον αφορά στις ε, μορφές αναφορών που συχνά λαμβάνετε στην Επιτροπή σας, θα ήθελα να πω ότι οι περιβαλλοντικές προσφυγές είναι οι περισσότερες ε, με βάση τους αριθμούς. Ε, όσον αφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι αλήθεια ότι υπάρχει έλλειψη πλήρης πληρο, πλήρους πληροφόρησης σχετικά με το ποια είναι τα δικαιώματα και τι μπορεί ο παρεμβαίνων αναφέρον να περιμένει από τα θεσμικά όργανα. Το πεδίο λοιπόν ε, των ε, δικαιωμάτων αυτών θα μπορούσε να γίνει καλύτερα κατανοητό αν εξηγηθεί καλύτερα από την Επιτροπή ε, μέσα από μία έκθεση τήσια για αυτό το θέμα. Επίσης, Όσον αφορά στη χάρτα, επειδή αυτή έχει μεταφερθεί ε, μέσω ευρωπαϊκού δικαίου, εμείς ε, ε, από την Κομισιόν δεν έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε. Όσον αφορά την αργοπορημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, τώρα με την συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να προτείνουμε κυρώσει μέσα από το δικαστήριο. Ε, πέρυσι, στο τέλος του έτους, ε, έγινε κάτι τέτοιο όταν η Κομισιόν ξεκίνησε τρεις ή τέσσερις τέτοιες υποθέσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν έχουμε ακόμα τις αποφάσεις του δικαστηρίου, όμως από τη στιγμή που δόθηκε η πρώτη ειδοποίηση, τα, μέσω της πρώτης επιστολής, τα κράτη-μέλη γρήγορα ξυπνούν και κάνουν κάτι. Έτσι λοιπόν, ε, κατά τις πρώτες μας εκτιμήσεις, ε, το εργαλείο που έχουμε μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας τελικά φαίνεται να δουλεύει. Όσον αφορά στο ρόλο των κρατών μελών, φυσικά παρεμβαίνουν αναφέρεται κατά της ε, διοίκησης. Να πω όμως ότι η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα επιτόπου έρευνας. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις γίνεται αυτό. Όχι κανονικά για μία κανονική προσφυγή. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας δίνει η συνθήκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν, σύμφωνα με τη συνθήκη, την ε, υποχρέωση συνεργασίας μαζί μας. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 και το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτό. Να αναφέρω επίσης ξεκάθαρα ότι οι αναφέροντες πάντοτε, ε, ε, οι καταγγέλλοντες πάντοτε ενημερώνονται πολύ συγκεκριμένα για κάθε στάδιο της διαδικασίας και αυτό επιβεβαιώνεται και με την ανακοίνωση που σας ε, απέστειλα το 2002. Την αναθεωρήσαμε πρόσφατα τον Φεβρουάριο ε, όπου επιβεβαιώθηκε αυτό ε, γιατί εξετάσαμε προσεκτικά και είδαμε ότι αυτό συμβαίνει. Ε, ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Το Σας ευχαριστώ για αυτή σας την παρέμβαση. Θα έχουμε συζήτηση για το όλο θέμα ξανά και με την ευκαιρία τη συζήτηση των τροπολογιών στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Γκέριγκερ, για την δουλειά να κλείσουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό και να δώσω το λόγο στους υπευθύνου για την διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία. Αυτή του Βερολίνου θα την συζητήσουμε το απόγευμα, όπω ζήτησε η συνάδελφο Λεποδά. Για την επίσκεψη λοιπόν στη Ρουμανία, νομίζω ότι πετύχαμε ένα σημείο ισορροπίας στο χρόνο που είχαμε από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Δεν υποβλήθηκαν, δεν πετάξαν αντιρρήσεις στο έγγραφο που σας υπέβαλα. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο μπορεί να θεωρείται εγκεκριμένο. Όπω διατυπώθηκε. Να δώσω το λόγο στου συνάδελφου που παρίστανται, εάν θέλουν να λάβουν το λόγο, ο συνάδελφο Μποστινάρου, για να συμπληρώσει κάποιε πληροφορίε. distinși colegi, raportul privitor la vizita... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση για την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών στη Ρουμανία έχει ως εξής. Επτά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, καθώς και ορισμένοι επιπροσθέτως Ρουμάνοι βουλευτές έλαβαν μέρος. όπου επισκεφθήκαμε στην Ρουμανία, παρά, αντίδραση, παρά την αντίδραση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχαμε πολλά ζητήματα στην ημερήσια διάταξη της ε, αποστολής μας. Προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν μια ιδηλιακή εικόνα της σημερινής καταστάσεως στη Ρουμανία. Ωστόσο, θα σας ευχαριστήσω πρώτα κυρία Πρόεδρε για τα εισαγωγικά σας λόγια και εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι το κείμενο που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ πιο ισορροπημένο και πολύ πιστότερο στην ρουμανική πραγματικότητα. Ανταποκρίνεται πολύ περισσότερο άλλωστε στις καταγγελίες των αναφερομένων. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών της χώρας. Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει όταν έγινε η ερευνητική αποστολή ότι σήμερα στην παρούσα επίσκεψη θα μπορούσαμε να δικαιωθούμε. Δηλαδή με την έννοια ότι τα πράγματα είναι όντως σημαντικά, ότι τα προβλήματα είναι σημαντικά, ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους Ρωμάνους πολίτες. Σήμερα ωστόσο επαληθεύεται η υπόθεση αυτή, διότι σήμερα λαμβάνει την υποστήριξη της Ρουμανικής Βουλής η νέα κυβέρνηση. Και έχουμε το θέμα των χρυσορυχείων στην Ρώσα Μοντάνα. Το έργο αυτό έχει ανασταλεί προσωρινά. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει τώρα σε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με, τις, με την κοινωνία των πολιτών, με τις μη κρατικές οργανώσεις, με, τις, με τους επιστήμονες και θα διερευνήσει κατά πόσον το έργο συμμορφώνεται με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τις σωρευτικές επιδράσεις της υλοποίησης του έργου. Θα εξετάσει επίσης κατά πόσο η οδηγία σε Βέζο, η οδηγία που λέγεται οδηγία σε Βέζο, γίνεται σεβαστή και κατά το πνεύμα της, αλλά και κατά το γράμμα της. Η επίσημη αυτή στάση της κυβερνήσεως, όπως εγκρίθηκε και από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο, δείχνει και πάλι ότι οι αναφερόμενοι είχαν δίκιο. Ότι οι Ρουμάνοι βουλευτές, αλλά και άλλοι από άλλες χώρες, οι οποίοι έφυξαν το θέμα, οι οποίοι, ε, ε, και, ότι και αυτοί δηλαδή δικαιώνονται και ότι είναι πραγματικές οι ανησυχίες τους και επιφυλάξεις τους. Και γι' αυτό χαίρομαι και για την θέση που λαμβάνει εν τέλει η έκθεση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές αξίες. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου, εγώ χθε είπα ήδη ότι προτίθεμαι να αποσύρω μια τροπολογία που ζητούσε κάτι απλό. Δηλαδή μια απλή προσθήκη. Ότι δηλαδή τέσσερα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τους αναφερομένους, οι οποίοι είχαν καταθέσει αναφορά για την ελευθερία του τύπου και ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αντέδρασε σφοδρά κατά της συζητήσεως του θέματος αυτού της ελευθερίας του τύπου, δηλαδή στη διάρκεια της επισκέψεως. Γνωρίζω ότι για ορισμένους εκτός συναδέλφων μου η ελευθερία του τύπου τους φαίνεται μάλλον βλαβερή για την υγεία του κόσμου. Ωστόσο, και γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε όλους και όλους ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Αυτό το έδειξε και αυτή η τελευταία Κυριακή. Αυτή η εντό εισαγωγικών Super Sunday. Πρόκειται για σημαντικές και βαθιές αλλαγές που επέρχονται. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση Πόντα που εγκαταστάθηκε τώρα θα διαγράψει από την εθνική τη στρατηγική, το τμήμα εκείνο που λέει ότι μπορεί να θυσιαστεί η ελευθερία του τύπου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ελπίζω δε και, άλλα, και άλλες πτυχές των πολιτικών ελευθεριών επίσης να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την έκθεση αυτή και ελπίζω πολύ να συζητηθεί και στι άλλε συναρμόδιες κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφου Και θέλω να είμαι βέβαιο ότι και οι πολίτες της χώρας μου, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτε στο σύνολό του, ελπίζω και εύχομαι να κατανοήσουν καλά ότι οι αξίε υπέρ των οποίων αγωνιζόμαστε καθημερινά και ιδίω εδώ στην δική μας Επιτροπή Αναφορών, όντως ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και συμφέροντα των πολιτών μας. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή και την κατανόηση που δείξατε απέναντί μας στη διάρκεια των τελευταίων μηνών όπου έγινε και η ερευνητική αποστολή της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών στη Ρουμανία. Όπως είπε ο κ. Μποστινάρου, η ερευνητική αυτή αποστολή κατέληξε να είναι πολύ περιπλοκότερη από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ο κ. Μποστινάρου απεφάσισε να αποσύρει την τροπολογία του. Μια τροπολογία η οποία δεν ήταν, δεν ε, αντιστοιχούσε σε κάποιο αντικείμενο της αντιπροσωπείας, της αποστολής μας. Αυτό δείχνει για μια ακόμη φορά ότι η Επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών εννοώ, Μπόρεσε έτσι να αποφύγει την εμπλοκή της σε παθιασμένες συζητήσεις και να λάβει το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς. Εμείς προσπαθούμε βέβαια, όντας αντιπολίτευση τώρα ε, στην νυν κυβέρνηση, να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Δεν θα αλλάξουμε βέβαια και τις απόψεις μας μόνο επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το κείμενο της εκθέσεως, έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Σε ανεπίσημες συζητήσεις αποφασίσαμε να εγκρίνουμε με συνένεση την έκθεση. Ελπίζω, ε, συγγνώμη, πιστεύω ότι όπως είναι τώρα η έκθεση, περιλαμβάνει ορισμένα θέματα που ακόμα δεν μπορούν να γίνουν πλήρως αντικείμενο συνενέσεως. Στη 13 για παράδειγμα. Το Κοινοβούλιο αποδέχεται λίγο πολύ την θέση των Ρουμανικών αρχών και αντιτίθεται έτσι στην αρχή της επικουρικότητας. Εγώ βρίσκω ότι θα ήταν λάθος να εγερθεί εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει αποφάσεις αντί των ρουμανικών αρχών. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μιλήσουμε για συστάσεις του Κοινοβουλίου. Και μιλώ για την σελίδα 13, παράγραφο 2. Να μην εγερθεί η εσφαλμένη εντύπωση στους ε, Ρουμάνους πολίτες ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω ο κ. Μποστινάρο να συμφωνήσει. Επίσης στην σελίδα 14 παράγραφο 2 όπου γίνεται παραπομπή στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου μας του Μαΐου του 2010 εδώ πάλι προκαλείται η εντύπωση ότι το ψήφισμα αυτό έχει κάπως διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα μη νομοθετικό κείμενο. Εγείρεται η εντύπωση ότι πρόκειται για νομοθετικό κείμενο. Δυστυχώς ο συνάδελφός μας, ο οποίος είχε τότε συντάξει προσθήκη στο κείμενο αυτό, προκαλεί με τον τρόπο αυτό την εντύπωση ότι η Κομισιόν θεσπίζει μια υποχρέωση. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Ο κ. Μποστινάρου μας έχει καλέσει κατ' επανάληψη να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των επιστημόνων και της πανεπιστημιακής κοινότητας στη Ρουμανία. Εγώ θα χαρώ. Να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση του Ρουμανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου. Το Δεκέμβριο του 2011 το Ελόγο Ινστιτούτο εξέδωσε γνωμοδότηση, η πραγματογνωμοσύνη θέλετε και έχω μπροστά μου και τα ρουμανικά και τα αγγλικά. Το κείμενο δηλαδή και στα ρουμανικά και στα αγγλικά και ευχαρίστω να το καταθέσω. Όπου ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου μετά από μελέτη που διεξήγαγε στην συγκεκριμένη περιοχή λέει καθαρά ναι για την υλοποίηση του έργου. Λέει δηλαδή ότι το Ρουμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο σας ενημερώνει ότι διεξήγαγε μελέτη επιπτώσεων για τις ενδεχόμενες δηλαδή περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και στη βάση της μελέτης αυτής τονίζει και πάλι την έγκρισή του για την υλοποίηση του έργου. Άρα το Γεωλογικό Ινστιτούτο έχει θεωρήσει ότι το έργο είναι χρήσιμο. Γιατί άραγε το κείμενο αυτό του Γεωργικού Ινστιτούτου να μην προσαρτηθεί στην έκθεσή μας για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να σας ζητήσω συγγνώμη και σε εσά και στην Επιτροπή γιατί έφτασα λίγο αργά. Ε, είχα καταλάβει ότι αυτό το θέμα θα συζητιόταν λίγο πιο αργά σήμερα το πρωί. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το έχω παρακολουθήσει. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις παρατηρήσεις του συναδέλφου κυρίου Πρέντερ με τις οποίες συμφωνώ. Είπε όμως ότι η η επίσκεψή μας ήταν λίγο πολύπλοκη στη Ρουμανία. Όχι, ε, δεν νομίζω ότι ήταν η επίσκεψη. Η, η κατάρτιση της έκθεσης έγινε λίγο περίπλοκη. Και γι' αυτό καταλαβαίνω γιατί ε, κάποιοι συνάδελφοι είχαν συγκεκριμένες απόψεις ε, παγιωμένες στην αρχή. Επίσης, να αναφέρω ένα σημείο που ανέφερε ο κύριος Πρέιντερ σχετικά με την έκθεση του Ρουμανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, γιατί ήδη έχει μιλήσει αυτός, αλλά στην ε, στο σχέδιο έκθεση, όπω το έχουμε ενώπιό μα αυτή τη στιγμή έχουμε όντω ένα παράρτημα, το παράρτημα 1 που έχει προσθεθεί μετά από την όλη εκδήλωση που είναι σημαντικό για το project. Ε, υποστηρίζω λοιπόν το αίτημα του κύριου Πρέντερ να συμπεριλάβουμε και αυτό το έγγραφο από το Γεωλογικό Ινστιτούτο στην έκθεση ουσιαστικά διότι καταρχάς έχουμε ένα προηγούμενο ε, με την προσθήκη μιας εξωτερικής έκθεσης ε, ε, μετά από το γεγονός κάτι που κάναμε με το παράδειγμα 1 και επίσης όταν έχουμε post factum εκθέσεις πρέπει να έχουμε μια ισόρροπη θεώρηση του θέματος. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια έκθεση που επικρίνει το project θα πρέπει να έχουμε και άλλη μία η οποία θα υποστηρίζει αυτό το project. Έτσι λοιπόν Ζητώ από την Πρόεδρο και την αντιπροσωπεία ε, της Επιτροπής ε, να εξετάσει ευνοϊκά το θέμα της προσθήκης αυτού του επιπλέον παραρτήματος στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Εφνερ. Ο κύριος Εφνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ερευνητική αποστολή στη Ρουμανία δεν ήταν απλή υπόθεση, νομίζω, για όλες και όλους μας. Ήδη διότι από την αρχή διεξήχθησαν πολλές και δύσκολες συζητήσεις για την κατάσταση της Ρουμανία στη βάση αναφορών που είχαμε λάβει, αλλά και επί τόπου δεν ήταν απλή η αποστολή αυτή. Χαίρομαι εν τέλει που για όλα τα βασικά θέματα μπορέσαμε να συνενέσουμε, μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και να δημιουργηθεί μια συνένεση για όλα τα βασικά θέματα λοιπόν της επισκέψεώς μας. Και κυρίως για το πιο κρίσιμο θέμα, δηλαδή την, ε, το έργο εξορίξεως χρυσού στην περιοχή Μοντάνα. Εγώ δεν προχώρησα στην επίσκεψη με προκατηλημένη άποψη. Προσπάθησα να ακούσω τις απόψεις όλων των πλευρών για να καταλήξω σε μια θέση. Εξάλλου δεν είναι δική μας υπόθεση της Επιτροπής Αναφορών δηλαδή να αποφασίσουμε τι θα κάνουν οι χώρες μέλη ή τι θα παραλείψουν, τι θα κάνουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ή τι θα παραλείψουν. Αυτό είναι όχι απλώς δικαίωμα της Ρωμανικής Κυβερνήσεως, είναι και σκόπιμο και προς το συμφέρον όλων μας να υπάρξει ανάπτυξη στη Ρουμανία που να αποδώσει τη θέμενη αξία και συνολικά στην Ευρώπη αλλά και στη Ρουμανία είναι χρήσιμο να αναπτυχθεί και η εξόριξη μεταλλευμάτων. Όμως όταν μας καλούν οι πολίτες να προσέξουμε, να εξετάσουμε εάν αραβιάζεται ενδεχομένω ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό ήταν το κύριο που με απασχόλησε εμένα στην αποστολή αυτή, δηλαδή να συμμορφούνται το έργο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να είναι βιώσιμο, να μην υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι είτε για τους ανθρώπους είτε για τη χλωρίδα και πανίδα. Αυτά ήταν σημαντικά για μένα. Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι στη Ρουμανία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό που ισχύει μέχρι τώρα, χρησιμοποιείται κιάνιο, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κιάνιο, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υδράργυρος, δηλαδή είναι τα πλέον επικίνδυνα τοξικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και σε ένα μέτρο και σε ποσότητες που δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Που προκαλούν λοιπόν σημαντικότατες βλάβες στο περιβάλλον και πάρα πολύ σημαντικούς κινδύνους για την υγεία του κόσμου. Εάν δηλαδή για παράδειγμα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν δηλαδή το κύκλωμα χρήσης των ουσιών αυτών δεν είναι απόλυτα ερμητικό. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που ακούω ότι η νέα ρουμανική κυβέρνηση επανεξετάζει σε βάθος τον σχεδιασμό αυτό και επιθυμεί να θέσει το θέμα ξανά και να το συζητήσει ξανά και να ανάλευει νέα απόφαση. Ελπίζω δε ότι και εμείς θα μπορέσουμε να εκφράσουμε την άποψη και τώρα και στο μέλλον ότι είμαστε μεν υπέρ της εξορίξεως ορυκτών μεταλλευμάτων και χρυσού βεβαίω, αλλά αυτό να γίνει σύμφωνα με την πιο πρόσφατη και ασφαλή για το κοινό τεχνολογία. Αυτά τα έχει πει σε ψηφίσματά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προετών, ειδικά για τη χρήση κιανίου για την εξόριξη χρυσού. Αυτά τα λένε άλλωστε και οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το δικό μα καθήκον. Και νομίζω αυτό πρέπει να αποτελέσει και διακομματικά τον στόχο μας. Υπάρχει και το θέμα το οποίο δυστυχώ λέω εγώ δεν αποτέλεσε αντικείμενο τη αποστολή μα. και το λέω δυστυχώ διότι είχαμε λάβει και σειρά επιγουσών αναφορών για το θέμα τη ελευθερία του τύπου στη Ρουμανία. Έχω τη μεγάλη ελπίδα τώρα μετά τις εκλογές και την εγκατάσταση της νέας κυβερνήσεως θα αντιμετωπιστούν σωστά οι δραστικές περικοπές της ελευθερίας του τύπου στην ε, ε, κατεπίκληση μιας νεφελώδους έννοιας της εθνικής ασφαλείας. Ελπίζω λοιπόν ότι και η δική μας Επιτροπή μπόρεσε και θα μπορέσει να συμβάλλει θετικά. Ευχαριστώ την εισηγήτρια καθώς και όλες και όλους τους ε, συμμετέχοντες για, την προσ... τις κοινές προσπάθειες, για μια ιστορία που δεν ήταν απλή και ελπίζω τα όσα είπα ως ελπίδες και ευχές να τα ακούσει και η νέα, Ευρωπα... Ε, η νέα Ρωμανική κυβέρνηση. Ο κύριος Πρώτον, ευχαριστώ την πρόεδρο της Επιτροπής που μπόρεσε να υποβάλει έκθεση που στο μεγάλο της μέρος βρίσκει τη συνένεση των βουλευτών. Ούτε και το περίμενα άλλωστε από την αρχή γιατί ήταν πολύ δύσκολο το θέμα. Δεύτερο, υπάρχουν ωστόσο επιθυμίες για ορισμένες τροπολογίες. Γι' αυτό θα ήθελα να ορίσουμε προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών και η ψηφοφορία της εκθέσεως να γίνει την επόμενη, στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν ξέρω πώ θα αντιμετωπιστούν διάφορες αυτές αλλαγέ. Απευθύνω έκκληση πάντω σε όλες και όλου. ναι με τροπολογίες αλλά να μην διαραγεί η συνένεση που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Η πρότασή μου πάντως είναι να γίνει η ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίαση. Ο κύριος Μποστινάρου, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας τώρα υποβάλλοντας νέες τροπολογίες. Αυτό θα καταστρέψει το περιεχόμενο της έκθεσης. Εάν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα έχει τέλος αυτή η διαδικασία. Δεύτερον, καμία δυνατότητα δεν υπάρχει να ε, προσθεθούν πληροφορίες, θα αποπείρει υπότιτε όχι, διότι έχει λήξει προθεσμία. Τρίτον, για το θέμα του ε, Γεωλογικού Ινστιτούτου. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρέντα που το ανέφερε, διότι ο πρώην διευθυντής, ο κύριος Μαρίντσα, απολύθηκε Ακριβώς γιατί ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος και ο υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής που αποτεμούσε το όλο εγχείρημα είχαν αντίρρηση με τις αρχές και τη φιλοσοφία του. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο απλώς και μόνο απολύθηκε και αντικαταστάθηκε. Όμως, με μία τελική απόφαση, ε, Ρουμανικό Δικαστήριο τις τελευταίες ημέρες, αποφάρθηκε, ο κύριος Στεφάν Μαρίντσα θα αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του ως Γενικός Διευθυντής του ε, Γεωλογικού Ινστιτούτου, οπότε θα βρίσκεται στη θέση του, θα φέρει εις πέρας το, πολιτικό του, το επιστημονικό του συγγνώμη, έργο χωρίς πολιτικές παρεμβολές. Τρία. Ένα εκ των υστέρων σχόλιο μετά από έπανε οι συνάδελφοι από χθε. Υπάρχει νέα κυβέρνηση με νέο πρόγραμμα. Εκεί ρητό αναφέρεται το πρόγραμμα. Ωραίο είναι να έχουμε φιλοσοφικέ και θεωρητικέ συζητήσει, όπω θέλετε πείτε τες, όμω στην πράξη νέα κυβέρνηση με νέο πρόγραμμα υπάρχει. Νέοι υπουργοί, όχι εκείνοι που συναντήσαμε κατά την επίσκεψη, που μα ε, έλεγαν πολλά ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί και έπειτα υπάρχει και τεχνική επιτροπή που θα ασχοληθεί με την όλη αξιολόγηση. Νέα λοιπόν πραγματικότητα, νέο πολιτικό τοπίο, νέα πολιτική βούληση. Ελπίζουμε ότι τώρα θα υπάρχουν ισόρροπες αποφάσεις και δίκαιε αποφάσεις από την ε, νέα κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την άριστη συνεργασία που είχαμε τους περισσότερους από τους συναδέλφους κατά την επίσκεψη αυτή και μετά την επίσκεψη. Αυτό τη συζήτησή μας θα πρέπει να την κλείσουμε κύριε Πρέντα. Ναι, ε, πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω σε αυτό που είπε και ο κύριος Γιάρ. Ε, συμφωνούμε. Συμφωνούμε και εμείς. Διότι υπάρχουν διαφορετικές πτυχές στην έκθεση αυτή. Αφορά μία επισκέψη που έχει ολοκληρωθεί. Μια επίσκεψη που ήδη έχει ε, γίνει λοιπόν, έχει δεξαχθεί και το κατά πόσο είναι φωτεινό ή όχι το μέλλον του σοσιαλισμού στη Ρουμανία. Θα το δούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της αντιπροσωπείας που συμμετείχαν σε αυτή την εσωτερική συζήτηση για την Ρουμανία. Ο κ. Ε, σας συγχαίρω προσωπικά διότι θεωρώ ότι αποτελεί προσωπική σας επιτυχία τη, ο συμβιβασμό στην έκθεση αυτή η οποία είχε τις ιδιαιτερότητέ της. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή δεν αφορά ε, παρά μόνον τα πορίσματα των ανθρώπων των, των μελών της Επιτροπής τα οποία επισκέφθησαν την ε, Ρουμανία και απεκόμισαν μετά από τη συζήτηση με τους διάφορους φορείς τα προσωπικά του συμπεράσματα. Έχω την εντύπωση ότι ε, από την παρούσα συζήτηση αντιλήφθηκα ότι ο κύριος Πρέντα προηγουμένως ήταν ε, υπέρ της προηγουμένης κυβερνήσεως και ο κύριος Μποστινάρου είναι υπέρ της παρούσης κυβερνήσεως. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι το θέμα, το είναι πιστεύω ότι υπάρχει, υπάρχουν ε, αναφέροντες σχετικά με ένα οικονομικό πρόγραμμα, την διεξαγωγή ενός επενδυτικού προγράμματος της Ρώσα Μοντάνα, το οποίο αποτελεί, ε, όπως είναι φυσικό, ε, θέμα που άπτεται τις αρμοδιότητες της ρουμανικής κυβερνήσεως και επομένως συνδέεται άμεσα με την αρχή της επικουρικότητας, και το οποίο ως φαίνεται είναι εκρεμές και ερχόμαστε υπό αυτού του θέματος προκαταβολικός πριν δοθούν οι άδειε και, έχουν, και έχει ολοκληρωθεί το θέμα να τοποθετηθούμε για παράβαση ή μη παράβαση κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, η άποψή μου είναι ότι η έκθεση όπως είναι έχει τις αναγκαίες αποστάσεις σχετικά με το θέμα Πιστεύω ότι η επένδυση, εγώ είμαι υπέρ των επενδύσεων γενικώ, φύση και θέση, διότι το μέλλον τη ανθρωπότητα και το οικονομικό μέλλον των λαών, ιδιαίτερα των τέως κομμουνιστικών χωρών, είναι με νέες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν εκεί για να δοθεί ε, μια κίνηση στην οικονομική ζωή των ε, κρατών. Α, έχω την εντύπωση ότι το Ρόζα Μοντάνα, αυτό είναι προσωπική άποψη που αποκόμισα από εκεί, είναι ότι αποτελεί ένα σχέδιο επένδυσης το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε στο μυαλό των επενδυτών από πλευράς οικονομικών μέσων υποστηρίξεως ε, με οικονομικά μέσα. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι η έκθεση ως έχει είναι ανώδυνη, είναι, τηρεί τις αναγκαίες αποστάσεις προς τις δύο απόψεις και έχω την εντύπωση ότι ε, πρέπει το ταχύτερο να περάσει, είναι δυνατόν και στην παρούσα συνεδρίαση διότι δεν κάνει τίποτε άλλο παρά τα πορίσματα, αναφέρει τα πορίσματα και περιγράφει τα πορίσματα των ανθρώπων που επισκεφθήκαμε την περιοχή εκεί. Και έχουμε κάθε απόψη, επειδή εγώ ήμουν ένα μέλος ε, από την Επιτροπή που ε, συνόδευα, είχα την τιμή να σε συνοδεύσω εκεί και τους άλλους κυρίους, ε, νομίζω ότι απηχεί το τι είδαμε και το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Το αν μελλοντικά το σχέδιο αυτό προωθηθεί από την κυβέρνηση που υπάρχει ή δεν προωθηθεί και αν παραβιάσει κοινοτικούς όρους ή δεν παραβιάσει θα το δούμε μελλοντικά. Προκαταβολικά πέραν της περιγραφής των όρων που είδαμε δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαλαβράκο. Ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς. Νομίζω είναι σαφές, όλοι συμφωνούμε, ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να εγκριθεί, όπως προτείνατε. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε κι άλλο για να υποβάλουμε τροπολογίες. Εγώ προσπάθησα να παρουσιάσω όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα τα γεγονότα όπω τα ζήσαμε. Γεγονότα που δεν έλαβαν αναγκαστικά πλαίσιο στο επίπεδο του επισήμου προγράμματος, αλλά περιλαμβάνουν όσα ζήσαμε και ακούσαμε. Σε ό,τι αφορά αλλαγές που θα θέλαμε να επέλθουν στο κείμενο, το κατά πόσο μπορεί να εμπλουτιστεί η έκθεση με κάποιες θέσεις ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση των θέσεων που εκφράζονται στο πρώτο παράρτημα της έκθεσης, εδώ θα ήθελα να παραμείνω συνεπής και εγώ με τα όσα έχω πει τώρα. Η θέση μου ως πρόεδρο της αντιπροσωπείας είναι ότι σε ένα τέτοιο έγγραφο δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κάτι το οποίο δεν ε, μας έχει γνωστοποιηθεί. Εδώ ζητήσαμε από όσους συμμετείχαν στο διήμερο, τρίμερο εργασιών που είχαμε εκεί, να τοποθετηθούν. Υπήρξαν συνάδελφοι που δεν είχαν χρόνο ομιλία, αλλά του ζητήθηκε να συμμετάσχουν στην εκπόνηση του εγγράφου. Με γραπτέ συνεισφορέ. Το έγγραφο που αναφέρει ο συνάδελφο Πρέντα Μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό υποβοηθητικό έγγραφο. Σας το έχει επισημάνει και η Προεδρία και προς ενημέρωση όλων θα μοιραστεί. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Αλλά δεν μπορεί να επισυναθεί στην έκθεση. Δεν είναι μέρος της αποστολή της επίσκεψης. Δεν συμπεριελήφθη στο πρόγραμμά μας τα όσα αναφέρει. μέρος λοιπόν του τεύχους ε, που καλύπτουν τις εργασίες μας θα μοιραστεί, θα διατεθεί σε όλους τους συναδέλφους που το επιθυμούν αλλά όχι κάτι παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα έλεγα ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή που θα ακολουθήσει την κανονική διαδικασία έγκρισης της ε, βάσει των αρμοδίτητων που πρόβλεπονται. Ο κύριος Γιάρ. Να πω ξεκάθαρα, αλλά δεν έχει να κάνει με το ταξίδι στη Ρουμανία, αλλά με την επίσημη ερώτηση. Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί έκθεση από συνάδελφα, εντάξει μπορούμε να το εγκρίνουμε, αλλά το θέμα είναι από τη δική μου πλευρά, από τη στιγμή που υπάρχουν τροπολογίες, πρέπει να ψηφίσουμε. Η αφελής ερώτησή μου λοιπόν είναι υπάρχουν τροπολογίες ή όχι. Αν δεν υπάρχουν, εντάξει. Αλλιώς θα πρέπει τουλάχιστον να ψηφίσουμε. Γιατί έτσι γίνεται ε, να λάβουμε απόφαση για αυτή την έκθεση στην Επιτροπή. Κύριε Γιάρ, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ακριβώς αυτό ήταν και το θέμα. Υπήρξε μόνο μια, ένα αίτημα να επισυναυτεί έγγραφο. Για αυτή την επισύναψη έδωσε όλη αυτή την απάντηση αμέσως πριν όπως και και ανάλογα αιτήματα που μπορούν να παρουσιαστούν. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Μα, κοιτάξτε, ίσως δεν ήμουν σαφής. Στη δεύτερη παράγραφο πρέπει να γίνει Αλλά Εγώ θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να προβάλλω τροπολογίες. δεν καλύπτεται επαρκώς το σημείο αυτό. Να μιλήσω για τη δική μου ομάδα. Εμείς ε, συμφωνούμε με την έκθεση ως έχει. Έχουμε κοπιωδώς ε, συζητήσει για αυτό το θέμα ε, πολύ καιρό και ε, ε, πραγματικά θα ήθελα να πω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι δεν θα μας άρεσε να έχουμε και πάλι τροπολογίες. Ε, δηλαδή δεν ήταν απλό να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω τι συμβαίνει, αλλά Εάν ε, δεν γίνεται να αποφασίσουμε, εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε για τις τροπολογίες σας, αλλά η δική μου θέση θα ήταν να γίνουν κάποια meetings με τους εμπλεκόμενους ε, και να συζητήσουμε έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε σήμερα να τελειώσουμε. Το άλλο θέμα είναι διάφορα έγγραφα τα οποία μπορούν να προσθεθούν αλλά δεν είναι κομμάτι της ίδιας της έκθεσης. Είναι πληροφορίες δηλαδή που προσκομίζονται. Αυτό ε, κατά τη γνώμη μου είναι εντάξει. Αν πρόκειται για το κείμενο αυτό αυτό ίσως θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε σήμερα έχοντας κάνει κάποιες συνεννοήσεις. Ο συνάδελφος ο κύριος Ποστινάρου. κυρία Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι άλλοι συναδελφοί μου, έτσι και εγώ έλαβα μέρος ε, στην σύνταξη των ε, τροπολογιών, τη συζητήσαμε εν μέρη με υποδύσκολους όρους και με μεγάλες εντάσεις συζητήσαμε. Υπήρξαν ε, κάποιες, κάποιες συμβιβασμοί, κάποια ευελιξία και οι διάφορες τροπολογίες και προτάσεις μπόρεσαν να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν από όλους. Ε, τελευταία, την περασμένη εβδομάδα εγώ προσωπικά ως ε, συντονιστής της ομάδας μου ανέφερα στους συναδέλφους ότι πρέπει να καταθέσουν τροπολογίες μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες τους απάντησα ότι ε, συμφωνώ με τις ε, συμβαστικές λύσεις μετά από τη συζήτηση στο Στρανσβούργο και συμφωνήσαμε όλοι ότι η έκθεση αυτή θα γίνει αποδεκτή, ε, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή υπό την παρούσα ε, μορφή. Ε, έχουμε λοιπόν εκπληρώσει όλες τις τυπικές διαδικασίες έτσι ώστε να μπορεί να εγκριθεί αυτή η έκθεση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που πραγματικά τηρήσατε ε, και λάβατε υπόψη σας όλες τις τυπικές διαδικασίες για αυτή την έκθεση. Στο μεταξύ, λοιπόν, θα έπρεπε να δώσουμε ένα τέλος ε, γιατί ε, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε αυτόν τον συμβιβασμό που καταφέραμε την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες προτάσεις. Αγαπητή ε, κυρία Πρόεδρε, ε, όντως είμαστε κοντά σε μία συμφωνία και θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που κάνατε και κάνατε πολύ καλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάποιοι ε, οι συνάδελφοι θέλουν ε, να εγκρίνουν την έκθεση ως έχει. Ο κύριος Μπρέντερ θέλει να καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Αν καταλαβαίνω σωστά την κοινοβουλευτική διαδικασία, αν δεν υπάρχει συμφωνία να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε όπως είναι η έκθεση, θα πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες και να ψηφίσουμε για αυτές το πού θα γίνει η διαπραγμάτευση, αν θα είναι στους διαδρόμους ή εδώ, δεν έχει σημασία. Πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες και να ψηφίσουμε μέσα στα πλαίσια της ε, τοπικής, τυπικής διαδικασίας όπως κάνουμε. Αν ο κύριος Μπρέγκερ ε, δεν θέλει να καταθέσει τις τροπολογίες, το ξεχνάμε και λέμε ότι υπήρξε ε, συνενετική λύση. Perfetto, se c'è ε, questa richiesta εφόσον υπάρχει τέτοιο αίτημα, πρέπει να ακολουθήσουμε και τον κανονισμό. Έλπιζα ότι θα απορροφηθεί τροποντινά το αίτημα αυτό, αλλά αναγκαστικά θα υποβληθούν τροπολογίες. Εγώ αρχικά δεν το είχα καταλάβει από τις πρώτες παρεμβάσεις. Σε αυτό το σημείο λοιπόν προτείνω την ίδια προθεσμία που προβλέφθηκε για το έγγραφο της επίσκεψης στο Βερολίνο. Παρασκευή το μεσημέρι. Ως τότε πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες και στην επόμενη συνεδρίαση θα ψηφίσουμε και για το έγγραφο και τις τροπολογίες. Ο συνάδελφος Έφνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν ακολουθήσουμε το αίτημα του κυρίου Πρέντα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά αυτό που, που εξηγήσατε εσείς. Με την ευκαιρία πάντως θα ήθελα να παρακαλέσω πραγματικά πολύ θερμά όλες και όλους τους συναδέλφους να σκεφτούν τι έχουμε επιτάπητος, διότι σπάνια έχω παρακολουθήσει τόσο δύσκολες διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Είχαμε μια deadline, όλοι γνώριζαν ότι μπορούσαν να καταθέσουν τροπολογίες, το κάναμε, καθίσαμε διαβουλευθήκαμε, καταλήξαμε σε μία λύση, κύριε Πρέντα, ακούστε με λίγο, που για την ώρα τουλάχιστον, επί της οποίας μάλλον για την ώρα, συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Φοβούμε ότι εάν αφαιρεθεί κάτι από αυτήν την ε, ε, θέση, θα αρχίσει πάλι η συζήτηση από την αρχή. Πραγματικά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε αν όντω είναι απαραίτητο να γίνει αυτό που προτείνετε. κύριος, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω είναι απλή η διαδικασία. Όμως κάποιες παρατηρήσεις δεν τις καταλαβαίνω. Ακούσαμε από τη σημερινή συζήτηση τι μας είπε ο κύριος Ποστινάρου. γιατί εκείνος να μπορεί να κάνει προτάσεις. Για παράδειγμα, ο κ. Μποστινάρου απέσυρε μια τροπολογία. Ωραία. Γιατί δεν δέχεστε λοιπόν και εμείς να έχουμε κάποιες τροπολογίε ή ενδεχομένω να αποσύρουμε κάποιες άλλε. Ας ισχύσει το ίδιο για όλους. Εάν ο κ. Μποστινάρου επιθυμεί να επιφέρει κάποιες αλλαγές, θέλω και εγώ να έχω το δικαίωμα να επιφέρω κάποιες αλλαγές, που ίσως μάλιστα είναι και πολύ σημαντικότερες από τις δικές του. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση, λέει η Πρόεδρος, για το θέμα αυτό ξανά. Μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες, ο κύριος Μποστινάρου. Κοιτάξτε, είναι γεγονός. Σας απέστειλα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ε, ε, μια φράση ότι δεν πρόκειται να καταθέσω τροπολογία για την ελευθεροτυπία μόνο και μόνο για να αποφύγουμε τη νέα διαδικασία, για να αποφύγουμε τις νέες εντάσεις και για το πολύ απλό γεγονός ότι κυρίως ήταν η δική σας εργασία αυτή που οδήγησε στην συνένεση. Και επειδή ακριβώς σέβομαι τη δουλειά σας και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρατε να υπάρξει συνένεση, γι' αυτό θεώρησα ότι είναι η πιο συνετή προσέγγιση από τη δική μου πλευρά και αυτό έκανα. Είναι, δεν είναι αναγκαίο να τροποποιήσουμε τίποτα στη δική σας εργασία. Ούτε χρειάζεται να υποψιάζονται τίποτα οι συνάδελφοί μου. Εγώ τάσομαι υπέρ της διατήρησης της συνενέσεως. Αν οι αξιότιμοι, μάλλον προς τους αξιότιμους συναδέλφους ε, του Λαϊκού Κόμματος. Ε, το μήνυμά μου είναι το εξή. Να ξανακαθίσουν να δουν, ή μάλλον τρεις οι συντονιστές έφτιαξαν την συνένεση, τη συμβαστική πρόταση. Θέλετε να ξανααρχίσουμε από την αρχή και τότε χάνουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε την έκθεση. Ή εν τέλει Ενδεχομένω να εγκριθεί μια διαφορετική έκθεση από αυτήν που έχετε υποβάλει εσεί, η οποία πέτυχε το συνένεση και να πάει χαμένη όλη αυτή η καλή δουλειά. Η δική μου έκκληση είναι να σεβαστούμε τους κανόνες και να μην επινοήσουμε νέους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους υφισταμένους δηλαδή βάσει των οποίων καταλήξαμε στην συνένεση αυτή, σε συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Εγώ ο ίδιος έχω μπει σε πολλούς αγώνες και σε πολλές διαμάχες. Αλλά ξέρετε και εσείς οι ίδια πόσο δύσκολο ήταν και πόσο οδυνηρό ήταν για ορισμένους από εμά να αποδεχθούμε κάποιες, ε, κάποιους συμβιβασμούς. Όμως αυτός είναι ο τρόπος. Διότι αλλιώς είναι περιτές διαμάχες οι οποίες μόνο ζημιά προκαλούν. Ευχαριστώ συνάδελφε Μποστινάρου. Όλοι έδειξαν την ανάλογη αφοσίωση αλλά εάν υπάρχει τέτοιο αίτημα δεν μπορώ να παρακάμψω τον ίδιο τον κανονισμό. Ορίζουμε λοιπόν την προθεσμία όπως προείπα. Σας ευχαριστώ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας ε, και το σεβασμό προς το άτομό μου. Όμως όλες οι συμπεριφορές είναι θέματα τακτικής που μας τα επιτρέπει και ο κανονισμός. Ο κύριος Γιάρ μπορεί να ζητά ψηφοφορία. Ζητήθηκε βάσει του κανονισμού και από άλλους συναδέλφους. Σε κάθε περίπτωση προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών Παρασκευή το μεσημέρι. Ελπίζω η ψηφοφορία να δώσει θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ όλους. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά και μετά αμέσω συνεχίζουμε με τι συνεδρίες των συντονιστών με 35 λεπτά καθυστέρηση.